Okay, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Εγκρίνεται? Καλώς, ευχαριστώ. Εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρίαση της 26 η Μαΐου και της 5 ης και 6 ης Κύριε Μπούρχερ για τα πρακτικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μια διόρθωση μάλλον που δεν ε, έχει γίνει. Αφορά τα πρακτικά της 26ης ε, Μαΐου στο σημείο 5 στην ψηφοφορία διαρθρωτικά μέτρα για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των ε, τραπεζικών ε, ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Εδώ πέρα το αποτέλεσμα είναι 21 ναι και 30 κατά και καμία αποχή. κυρία Πίτη Κάινεν δήλωσε απέναντι στην γραμματεία πως δεν λειτουργούσε το μηχάνημά της και είχε άρα ψηφίσει ναι, είναι 30-30 λοιπόν το οποίο δεν αλλάζει τίποτα στο αποτέλεσμα πάλι απορρίπτεται αλλά νομίζω θα πρέπει να καταγραφεί σωστά στα πρακτικά. Έτσι. Απλά ήθελα να το παρατηρήσω. I, I can, uh, Ναι, εκτός και αν θέλετε το λόγο μπορώ να απαντήσω. Καλώς. Έλαβα την επιστολή της κυρίας Κάινεν και βεβαίως σημειώνουμε την ε, αποστολή της επιστολής και μπορούμε να κάνουμε αναφορά στα πρακτικά, αλλά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αλλάξουν αναδρομικά. Και εξ όσων αντιλαμβάνομαι, έχει καταγραφεί η ψήφος. Ψήφισε η κυρία Πιετικάνεν. Ίσως ήταν τεχνικό το λάθος αλλά ήταν ηλεκτρονική η ψηφοφορία και ο αριθμός που είχαμε συμπεριλάβει ήταν αυτός της κυρίας Πιετικάινεν. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Σημειώνω την ύπαρξη της επιστολής, της εμπεριλαμβάνω στα πρακτικά, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και προσοχή ε, θα άλλαζα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και άλλωστε δεν αλλάζει και η ουσία. Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα και ένα νομικό ζήτημα. Σε αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πρέπει να διαβουλευθώ με τους ειδικού. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε την έγκριση των πρακτικών υπό αίρεση και να κάνουμε την κατάλληλη διαβούλευση με τις τεχνικές και νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποια είναι η συνήθις διαδικασία υπό αυτές τις συνθήκες. Ελίζα. Ναι, γι' αυτό το ζήτημα ήθελα να μιλήσω και εγώ ήμουνα παρούσα στην ψηφοφορία και δεν θυμάμαι να έγιναν εκ των προτέρων ανακοινώσει. Συχνά το κάνουμε και λέμε ότι το μηχάνημά μου για την ψηφοφορία δεν δουλεύει, η κάρτα δεν μπαίνει κτλ. Επομένως, Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε, δεν μίλησε κανείς για τεχνικό πρόβλημα, μπορεί κανείς να στείλει επιστολή, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά κριτήρια από τη μία συνεδρίαση στην άλλη. Ο Πρόεδρος. Καλώς, σας μείνουμε εδώ σε αυτό το θέμα και επανερχόμαστε. Δηλαδή η έγκριση των πρακτικών είναι υποαίρεση, θα, θα τα εγκρίνουμε αύριο ή στην επόμενη συνεδρίαση και πριν περάσουμε στα σημεία 3 και 4 και 5 της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να πω στους συναδέλφους κάτι για τη συνάντηση της συνεδρίασης των συντονιστών. Έγινε ένα αίτημα και θα τροποποιήσουμε ελαφρά τη διαδικασία μας ως προς το χρόνο που έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Θα πάμε σε ένα αυτόματο σύστημα όπου το μικρόφωνο θα κλείνει μετά το πέρας του χρόνου που έχει ε, το κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάθεσή του. Θα δούμε πώς δουλεύει το σύστημα, θα ε, ξεκινήσω από σήμερα και θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους, να το κάνετε και εσείς, ότι δηλαδή ε, πέντε λεπτά έχει ο καθένας στη διάθεσή του, στο τέλος των πέντε λεπτών θα το κλείνετε το μικρόφωνο, θα κλείνει το μικρόφωνο του. Θα ζητήσω λοιπόν από τους συντονιστές να θέσουν σε ισχύ αυτή την απόφαση αναλόγως και θα ζητήσω από τους συντονιστές να ζητήσουν από τους συναδέλφους να φτάνουν έγκαιρα ή πρέπει να ξεκινούμε τη συνεδρίαση χωρίς την παρουσία ε, των απαιτούμενων συναδέλφων και αυτό δεν είναι καλό. Περνάμε λοιπόν στα σημεία 3, 4 και 5 διάταξης. Μιλούμε για την ακρόαση με τους τρεις προέδρους των τριών ΕΖΑΣ είναι μια ακρόαση που συνάδει με το άρθρο 51 του κανονισμού ΕΖΑΣ αλλά δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση για εμάς να έχουμε μια τέτοια ακρόαση, αλλά είναι και χαρά, διότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τους τρεις. Φυσικά, σε κάθε συνεργασία υπάρχουν θέματα πάνω στα οποία διαφωνούμε, πάνω στα οποία συμφωνούμε. Ε, μπορεί να υπάρχουν θέματα που επιδέχονται βελτίωση, σίγουρα. Εγώ προσωπικά όμως είμαι πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία μας με τους ε, τρεις ε, προέδρους της ΕΖΑΣ. Σας καλωσορίζω επισήμως και χαίρομαι διότι έχουμε αυτή τη συνάντηση και θα ε, βάση της νομική που, που, που εξαρτάται από τη νομική μας βάση ε, πρέπει να εξετάσουμε την περασμένη χρονιά αλλά και τις εξελίξεις στο μέλλον είναι κρίσιμη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει ε, το Single Rule Book η εντολή για ενιαίους κανόνες φαντάζομαι ότι και οι τρεις πρόεδροι θα αναφερθούν σε όλα αυτά τα θέματα Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Στίβεν Μάιτζορ, πρόεδρο ο οποίος θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του. Μετά ο κύριος Ανδρέα Ενρία και ο κύριος Γκάμπριελ Μπερναρτίνο θα έχουν από 5 λεπτά και μετά θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές και θα τους κλείσουμε το μικρόφωνο μόλις τελειώσει ε, ο χρόνος τους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο, για την εισαγωγή σας και τις θετικές παρατηρήσεις για την συνεργασία μεταξύ ΕΚΟΝ και ΙΕΖΑΣ και βεβαίω είναι αμοιβαία τα αισθήματα, θα έλεγα. Άκουσα πως θα είστε πάρα πολύ αυστηρός να με το χρόνο να μπούμε λοιπόν, λοιπόν απευθείας στην ουσία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Κυρίες ε, και κύριοι, το 2015 η Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών είναι επικεφαλής ε, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και ως πρόεδρος της ενικτής Επιτροπής θα ήθελα να αναφέρω τις ε, κυριότερες δραστηριότητες μας το τελευταίο έτος. Η κοινή αυτή επιτροπή λειτουργεί ως το φόρουμ συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών ε, κινητών αξιών και αγορών. Θα ήθελα να πω πως ε, επικεντρωνόμαστε στην προστασία του καταναλωτή και στο να διαπιστώνουμε και να αξιολογούμε που υπάρχει διατομεακός κίνδυνος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο μη εκείνους ε, που απαιτούν συνεργασία στους κλάδους της αγοράς, των ασφαλιών και της τράπεζας μεταξύ των οποίων και η κεφαλαιοποίηση και η τηλεοποίηση και η χρηματοοικονομική όμιλη. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ κυρίω στην κοινή εντολή για τα τρίψο που έχουμε δημοσιεύσει δύο έγγραφα εργασία και θα δημοσιεύσουμε άλλο ένα το Νοέμβριο. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε πω με τα έγγραφα αυτά οι καταναλωτέ λιανική θα μπορούν να αντιληφθούν και να συγκρίνουν επενδυτικά ε, και ασφαλιστικά προϊόντα. Επιπλέον, ε, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ για τις πρακτικές ε, πολλαπλών απολύσεων και κοιτάμε να δούμε επίση τι γίνεται στον τομέα των χρηματοοικονομικών συμβουλών σε καταναλωτέ λιανικής και κοιτάμε επίση. Ε, είχαμε και μια ημερίδα στην Φραγκφούρτη για το θέμα αυτό που μα έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε με του εκπροσώπου των καταναλωτών. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα την ε, κοινή και διαδομαϊκή αξιολόγηση κινδύνου, συντάξαμε δύο εκθέσεις ε, που εστιάστηκαν στην ταυτοποίηση κινδύνων ε, και ασθενών σημείων στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική κίνδυνη λοιπόν είναι η ασθενής οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης, ε, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, η μεγάλη κινητικότητα στις αγορές και η χαμηλή κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επιπλέον. Η Κοινή Επιτροπή αξιολόγησε τους κινδύνους όσον αφορά την διεξαγωγή των ε, επιχειρήσεων στους ε, κλάδους ε, των ασφαλιών και των τραπεζών. Τέλος, όσον αφορά τις συστάσεις μας, δύο έντολες σύμφωνα με την οδηγία για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2014 και έχουμε προετοιμάσει σχέδια κοινών τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τους κανονισμούς για την κεφαλαιακή επάρκεια και την τα 2 όσον αφορά επίσης ε, και την ε, μεταρρύθμιση της ε, οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μία αναβίωση των αγορών τιτλοποίησης στην Ένωση και εκεί πέρα ακριβώς εντοπίσαμε τα κενά και τις ασάφειες που υπάρχουν στο αριθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης και το που υπάρχουν διάφορες Αναγνωρίζοντας βεβαίως όλες τις καλές προσπάθειες της ΕΚΟΝ για να βελτιωθεί ο προπολογισμό μας, θα ήθελα να σημειώσω πως φέτος εργαζόμαστε με πόρους που είναι κάτω από το απαραίτητο επίπεδο για να επιτύχουμε αυτά που μας έχουν ανατεθεί. Το σχέδιο προπολογισμού για το 2016 δεν βελτιώνει και σε κάποιες περιπτώσεις επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση των αρχών χωρίς ε, να αν δεν επανεξεταστούν αυτά τα πράγματα θα αναγκαστούμε να καθυστερήσουμε στην επίτευξη των παραδοτέων. Τέλος, να πω πως ε, και το επόμενο έτος θα συνεχίσουμε να ε, συνεργαζόμαστε και βεβαίως αυτό έχει κέρια σημασία, συνεργασία δηλαδή μεταξύ των αρχών. Θέλουμε η συνεργασία μας να είναι στο δυνατόν πιο διαφανής, να σεβόμαστε αυτά τα οποία έχουν χαρακτήριος ω ε, κανόνες και να ενταθεί και η άτυπη ανταλλαγή απόψεων. Και βεβαίως θα σα υποβάλουμε γραπτός ε, και προφορικός αναφορές ε, για τις επιλογές που σκοπεύουμε να κάνουμε και για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Τώρα να περάσω στο κομμάτι που αφορά την ΕΣΜΑ. Για να σας παρουσιάσω την δουλειά της και τα επιτεύγματά τη στο προηγούμενο έτος. Βεβαίως γι' αυτό πρέπει αυτό να συνδεθεί με τους στόχους μας. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν δημιούργησε την ΕΣΜΑ για να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών και να διασφαλίσει την σταθερότητα και τη σωστή λειτουργία των χρηματαγώνων. Αυτό Αυτούς τους στόχους επιτυχάνουμε με δύο τρόπους, με το να, υπάρχει, να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες ε, για τις ε, κεφάλαια αγορές και να υπάρχει και ενιαία εφαρμογή τους, είτε μέσω της ρυθμιστικής σύγκλησης, είτε μέσω της απευθείας εποπτείας ε, των αποθετηρίων και των υπηρεσιών και οίκων Το προηγούμενο έτος λοιπόν εκδώσαμε πάνω από 100 σχέδια τεχνικών προδιαγραφών και όλα αυτά συνεισέφεραν στην μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, κεφάλαια αγορές, ε, κάτι το οποίο βεβαίως διατρέχει όλο το έργο μας επίπεδου 2, μεταξύ των οποίων MIFI2, MIFIR, EMIR, και CSDR. Όλοι αυτοί είναι οι κανονισμοί τους οποίους εφαρμόζουμε. Όταν λοιπόν χαράσουμε αυτούς τους ε, κανόνες, κοιτάμε να αντιμετωπίσουμε την ε, ασυμμετρία πληροφοριών για να μπορούν οι επενδυτές να κάνουν καλύτερες επιλογές αλλά και οι υποπτικές αρχές να επιτελούν το έργο τους. Πρέπει λοιπόν πριν εκπαιδεύσουμε νέους κανόνες να δούμε το κόστος και το όφελος και να τα ζυγίσουμε καθώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ε, κεφάλαια αγορές. Παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις απαιτήσει διαφάνειας έχουμε σε συνεργασία με, τους, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές καταλήξει σε ένα πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, για την συνεισφορά της σε αυτό το θέμα όπως και σε άλλα σημαντικά θέματα για το ΜΥΦΙΡ και θα διασφαλίσω πως οι διαβουλεύσεις μας στο Διοικητικό Συμβούλιο στα τέλη του μήνα θα τα λάβουν όλα αυτά υπόψη η διαβούλευση είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χάραξη κανόνων της ε, ΕΣΜΑ. Κάνουμε εντατικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και δίνουμε την ευκαιρία μέσω διαφόρων διάβλων για να μας δώσουν τις απόψεις τους. Επιπλέον, πέραν από τα μέτρα τεχνικής εφαρμογής, οι κανόνες αυτοί έχουν συνεισφέρει σε ευρύτερα ζητήματα όπως την βελτίωση των διάβλων χρηματοδότηση ε, των κεφαλαίων τη Ένωση. Έχουμε δώσει συμβουλέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το crowdfunding, την ε, τίτλοποίηση και τα ευρωπαϊκά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Επίση ε, συνεισφέραμε στην ευρύτερη συζήτηση για το CMU και για το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τι πιστοτικές πληροφορίε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τη διασυνοριακή λειτουργία του. Οι ενιαίοι αυτοί κανόνες λοιπόν μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε από νωρίς ε, που υπάρχουν ε, ζητήματα στα οποία απαιτείται ενιαία εφαρμογή για την ΜΥΦΙΡ. Έχουμε δει λοιπόν πως υπάρχει ανάγκη για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα συνδυάζει πληροφορίες από 300 σημεία στα οποία γίνονται συναλλαγές και όλες αυτές τις πληροφορίες να συγκεντρώνονται σε ένα όλα αυτά για να στηριξούμε την ενιαία αγορά. Όπως είπα, μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά απαιτεί και ενιαίους κανόνες αλλά και ε, ενιαίες, ε, ενιαία εποπτεία. Οπότε προσπαθούμε να οδηγηθούμε σε μια ρυθμιστική σύγκληση. Εργαζόμαστε λοιπόν σε κάποιες ε, αξιολογήσεις από ομοτήμους για να δούμε το trading υψηλών συχνοτήτων και βεβαίως τις ε, δίκες και παραπλανητικές ε, πληροφορίες για τους καταναλωτές. Επίσης, ε, φροντίζουμε οι ρυθμιστικέ αρχές να πηγαίνουν επί τόπου στους εποπτευόμενους και πέρα από όλα αυτά χρησιμοποιούμε και κάποια εργαλεία τα οποία απαιτούν λιγότερους ανθρώπινους πόρους όπως ερωτηματολόγια. Τώρα θα στραφώ στον, στον εποπτικό μας ρόλο, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την σταθερή λειτουργία των κεφαλαίων αγορών έχουμε οδηγηθεί έτσι όσον αφορά την σύρεση σε μεγαλύτερη σταθερότητα. Εξακολουθούμε να ψάχνουμε τομεί για βελτίωση. Παραδείγματο χάρη η ΕΣΜΑ επέβαλε για πρώτη φορά σε εποπτευόμενο οργανισμό το πρώτο της ε, πρόστιμο για προβλήματα στον εσωτερικό έλεγχο. Έχουμε λοιπόν ή μάλλον πλησιάζουμε περισσότερο προς μία ενιαία αγορά και μία ένωση παραγόγων. Η διαφάνεια βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ βασική για να έχουμε μια ασφαλή αγορά παραγωγών και εδώ πέρα εξακολουθούμε να ασκούμε τον υποτικό μας ρόλο. Το 2016 λοιπόν θα είμαστε 5 ετών και μέχρι τότε θα έχουμε ολοκληρώσει τον κύριο όγκο του έργου μας. Και περνάμε άρα στο πεδίο της εφαρμογής. Θα αφιερώσουμε περισσότερους πόρους στην ρυθμιστική σύγκληση και θα απομακρυνθούμε από το γράψιμο των κανόνων τέρος. Να αναφερθώ στην ε, Ένωση Κεφάλαια Αγορών. Είχαν πρώτα απ' όλα την ε, αντίδραση ε, στην οικονομική κρίση η οποία πήγαινε προς την κατεύθυνση της καλύτερης και πιο ενιαίας ρύθμισης κάτι το οποίο βεβαίω θα αποτελέσει ένα σημαντικό στατικό στοιχείο της ε, Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως είναι ε, ρυθμιστική αρχή βασικός παράγοντας για την οικοδόμηση της ε, ε, κεφαλαίου αγοράς. Και σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε λάβατε υπόψη και τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για αυτή την εισήγηση που σίγουρα είναι θετική προσέγγιση προς ε, τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ενερία που είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη αυτής της Επιτροπής έχει γίνει μεγάλη ε, πρόοδος όσον αφορά την οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομεριών των τραπεζικών μεταρρυθμίσεων όπως αυτές προβλέπονται στην οδηγία περί απαιτήσεων και ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών. Έχουμε γκρίνει 158 σε προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές και υπόλοιπα 117 προϊόντα που πρέπει να μας δώσει τραπεζική, μάλλον να εκδώσει η τραπεζική αρχή έχουν ήδη δοθεί στη δημόσια διαβούλευση και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί τις αρχές του 2017. Η εστίαση της EBA σταδιακά από το σχεδιασμό θα μεταβεί στην πραγματική και συνεπή εφαρμογή το, από πλευράς των εποπτικών αρχών της Ένωσης, καθώς και παρακολούθηση των δομών των αγορών, των πρακτικών των επιχειρήσεων, καθώς και την ποιότητα και την τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες στους πελάτες τους. Άρα ρυθμιστικά θέματα όπως οι, πληρω... υπηρεσίες πληρωμών σιγά σιγά αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στη δική μας ατζέντα. Είμαι ε, για την εξισορρόπηση ε, και τη σημασία του ενιαίου εγχειριδίου. Όμως η ανταπόκριση των τραπεζών θα εξαρτηθεί από την, ε, ε, το κατά πόσο θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ε, την ε, εξέλιξη και αυτό μπορεί να βασιστεί στην ολοκληρωμένη έκθεση που έχει και αναθεώρηση που έχει ανακοινώσει πρόσφατα η Κομισιόν. Προσωπικά πιστεύω ότι υπερβολικά λεπτομέρειες περιλαμβάνονται σε νομοθεσία επίπεδο 1 και μετά από τις αποφάσεις του 10 θα ήταν σωστό σε ορισμένους πολυτεχνικούς τομείς να αναθέσουμε περισσότερες ε, ευθύνε στην τραπεζική αρχή. Ένα παράδειγμα είναι η εποπτική έκθεση όπου πολύ συχνά είναι εξαιρετικά περίπλοκα τα όσα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα. Πρόσφατη εργασία της ε, EBA, της ε, Τραπεζικής Αρχής, έχει βασιστεί στον έλεγχο των εγγυήσεων όπως ε, το MRL, e δηλαδή τα διαθέσιμα και επίση έχουμε ξεκινήσει πολύ στερεί βάσει όμω οι καθυστερήσει στην εφαρμογή τη οδηγία ε, περί ανάκαμψη και εξυγένση των τραπεζών οδηγεί σε μια επιπλοκή. Γιατί όλε οι αρχέ δεν έχουν, όλα τα κράτη δεν έχουν ορίσει εθνικέ ε, ε, αρχέ εξυγίανση και γι' αυτό ε, και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την εξυγίαση πολύ συγκεκριμένα στις χώρες αυτές. Η εργασία μας για την τυπλοποίηση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μια ομοιόμορφη προσέγγιση βλάπτει την αγορά για, αυτές τις, ε, για, τα σχετικά ασφαλή προϊόντα τυπλοποίησης και πρόσφατα στις συμβουλές μας προς την Κομισιόν συστήσαμε να ληφθεί μια απόφαση στο αριθμιστικό πλαίσιο η οποία να ρυθμίζει τα, τα θέματα όπου οι εγγυήσεις θα ακολουθούν διαφορετικές δομές σε σχέση με τις ε, ε, με τους ίδιους πόρους της κάθε ε, εταιρείας ή της κάθε τράπεζας. Οι εκθέσεις που σας δίνουμε από το 2009 παρέχουν μία ανάλυση επί των γεγονότων όσον αφορά την επίπτωση στις μικρές επιχειρήσεις και στο δανεισμό για το σύνολο της οικονομίας. Πρόσφατες ε, έρευνες για τις ε, συστημικές ε, τράπεζες και την δυνατότητα απορρόφησης πλήρους ε, της πλήρους ζημίας μπορεί να οδηγήσει στην, σε κάποιες προσαρμογές. Όμως οι προποτινόμενες αλλαγές σε μεγάλο βαθμό είναι συμβατές με τις προδιαγραφές της ε, τραπεζικής αρχής. Θέλουμε να υπάρχει συνοχή και στις ε, απαιτήσει σε σχέση με τα ευαίσθητα σε κινδύνους κεφάλαια. Εμείς έχουμε λάβει επικοδομητικό ε, Επικοδομητικέ απαντήσει στη διάρκεια τη δημόσιας διαβούλευση, θα μπορέσετε να δείτε και έναν δικό χάρτη και εντατικοποιούμε τις προσπάθειε μα όσον αφορά την ε, σύγκριση επιδόσεων για τις ε, σταθμισμένους, για τους σταθμισμένους κινδύνους. Έχουμε επίσης ποδώσει μεγάλη προσοχή στην σωστή εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και τώρα οξύνουμε την προσέγγιση μας, ας πούμε, όσον αφορά την εξυγίανση και την ανάκαμψη. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στον τομέα των αμοιβών οδηγεί σε νομικά θέματα και κατά την γνώμη μας απαιτεί αλλαγές στο κείμενο επίπεδου 1. Επίσης προχωράμε με την ε, ατζέντα ε, που αφορά την ε, σύγκληση στην εποπτεία, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την ενιαία αγορά ε, και για την ε, Τραπεζική Ένωση. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα για τους επόπτες. Όπως ξέρετε, φέτος αποφασίσαμε να μην κάνουμε ε, τεστ αντοχής, αλλά διατηρούμε ε, τη δέσμευσή μας για μια εκτεταμένη προσπάθεια διαφάνειας που θα ολοκληρωθεί μας στα τέλη του χρόνου. Εν τω μεταξύ, ε, σχεδιάζουμε το, το τεστ για την προέλευση των, των κονδυλίων κάθε φορά και αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επίσης του χρόνου. Σε σχέση τώρα με την γνωμοδότησή μας για τα εικονικά νομίσματα, έχουμε εκδώσει μια σχετική γνωμοδότηση όσον αφορά την χρηματοδότηση από τον κόσμο, το crowdfunding, καθώς και οδηγίες σχετικά με ίδιες πρωτοβουλίες που αφορά την ασφάλεια στις πληρωμές στο ίντερνετ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, κύριε Ενερία. Πολύ πλούσια η εισήγησή σας. Και τώρα ο Γκαμπριέλ Μπερναρντίνο από την ΑΙΟΠΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να μοιραστώ μαζί σας τα επιτέματα αλλά και τις προκλήσεις για την ΕΙΟΠΑ. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η εποπτεία της σύγκλησης εμείς, ανέκα, εμείς ε, αυτό κάνουμε από τα τέλη του 2014 για να υπάρχει βέλτιστη δυνατή συνέπεια μεταξύ ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του Solvency 2. Και υπ' αυτή την έννοια έχουμε 18 εφαρμοστικά τεχνικά ε, πρότυπα, έχουν εναρμονιστεί οι προϋποθέσεις για το reporting και έχουμε δύο σετ οδηγιών που καλύπτουν τα περισσότερα θέματα του Solvency 2. Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές έχουν να κάνουν με την ευθυγράμμιση των βασικών διαδικασιών εποπτείας, αλλά άλλες παρέχουν μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις προσδοκίες ε, των εποπτών και μειώνεται ο κίνδυνος ε, η κάθε εθνική αρχή να δίνει τη δική της ερμηνεία. Εμείς ε, θελήσαμε να έχουμε μια πιο συνολική και λεπτομερή εικόνα των μεγάλων έργων υποδομής. Κάναμε ε, διαβούλευση τον Ιούλιο και είχαμε νέους ορισμούς, νέα κριτήρια έτσι ώστε να τύχει πιο ειδική μεταχείριση στο στάνταρ έντυπο που συμπληρώνεται ένα μεγάλο έργο υποδομής που έχει ίδια κεφάλαια και συμμετοχή του δημοσίου. Έχουμε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία υπάρχει στα template τα κανονιστικά του Solvency 2, στα βασικά πρότυπα. Επομένως, οι απαιτήσει ε, αναφοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ μειωμένες. Και για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο, το καλοκαίρι δημοσίευσαμε ένα εργαλείο ε, που θα τις βοηθήσει να δημιουργήσουν να επικυρώσουν και να επεξεργαστούν ε, έγγραφα εργασίας XML. Και θα το χρησιμοποιήσουν αυτό πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς την εφαρμογή δημοσιεύσαμε τα κριτήρια για το κίνδυνο και είχαμε εσωτερικά ε, μοντέλα εγκρίσεων. Τον Απρίλιο εκδώσαμε μια γνωμοδότηση για τα εσωτερικά μοντέλα και καλύψαμε εκεί την ε, έκθεση των κρατών αλλά και την ε, προσέγγιση των εποπτών και τις, αντι... τις διαδικασίες και αντιστοιχίας. Οι εθνικές αρχές έχουν ένα ανεξάρτητο feedback αντικειμενικό για την εποπτεία. Η ομάδα ήρθε σε έκανε 18 διμερείς επισκέψεις σε εθνικές αρχές και δώσαμε προσοχή στη συνεργασία με τη Ρουμανία για να ενισχυθεί η εποπτεία του τομέα εκεί. Κάναμε αναθεώρηση και κάναμε τα stress test, τα τεστ αντοχής των ασφαλιστικών εταιριών στην αγορά της Ρουμανίας και βρήκαμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές ε, στους ισολογισμούς και διάφορα άλλα στοιχεία και όλα αυτά τα μέτρα υιοθετήθηκαν. Ήταν μια αξιόπιστη άσκηση και αυτή ήταν θεμελιώδης για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή και εμπιστοσύνη στο τομέα των ασφαλιστικών της Ρουμανίας. Βεβαίως δουλέψαμε και πάνω στα διεθνή πρότυπα. Είμαστε παρόντες ε, σε διεθνείς φορείς και διεθνείς οργανισμούς και έτσι εκπροσωπούνται καλύτερα οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Έρχομαι τώρα στην προστασία του καταναλωτή, που είναι μέρος του DNA μας άλλωστε και το έχουμε πάντοτε ως προτεραιότητα. Έχουμε τη νέα οδηγία για την ασφάλιση των προϊόντων τη γνωστή και με αυτό είναι ο, γνώμος, ο γνώμονάς μας. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για την εποπτεία των επιχειρήσεων, ένα πλαίσιο που θα προβλέπει ε, το, τη βλάβη που μπορεί να υποστεί ο καταναλωτής και που δεν θα αντιδρά μόνο στη βλάβη που έχει υποστεί ο καταναλωτής, που δεν θα αντιδρά εκ των υστέρων. Έχουμε θεματικές επαναξιολογήσεις με δείκτες που θα ε, αξιολογούν και τον κίνδυνο και από πλευρά συντάξεων έχουμε τα ατομικά συντοξιδωτικά προϊόντα. Τον Ιούλιο κάναμε διαβούλευση, προτείναμε τη δημιουργία ενός προϊόντος ε, πανευρωπαϊκού για τις συντάξεις, το οποίο είναι αξιόπιστο και έγκυρο και αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ε, Ένωση Κεφαλαιογορών στην Ευρώπη. Βεβαίως Σύμφωνα με την εντολή που μας είχε δοθεί, συνεχίσαμε στο συντονισμό των τεστ αντοχής για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το ολοκληρώσαμε αυτό ε, το καλοκαίρι με βάση τις απαιτήσεις του Solvency 2. Δείχνουν τα τεστ ε, ε, αντοχής ότι ο ασφαλιστικός τομέας είναι σε κίνδυνο διπλάσιο από τα ίδια κεφάλαια και αυτό έχει να κάνει και με τα επιτόκια και με ε, τις προβλέψεις. Υπάρχει, είναι λοιπόν ευπαθής, εντοπίσαμε τα σημεία τα αδύναμα και ε, υποβάλαμε προτάσεις. Το Μάιο κάναμε τεστ αντοχής για τις ε, συντάξεις τις εργασιακές. Το πρώτο τεστ που έγινε στην Ευρώπη και είδαμε ότι πολλά από αυτά τα ταμεία είναι ευπαθή λόγω της ε, πτώσης των τιμών των στοιχείων ενεργητικού, όπως και στο, με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Προσπαθήσαμε να έχουμε διαφορετικές εποπτικές προσεγγίσεις για να βρούμε τη βέλτιστη και θα εκδώσουμε γνωμοδότηση για πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αξιολογείται το κατά πόσο είναι βιώσιμες οι συνταξιοδοτικές υποσχέσεις. Έρχομαι τώρα σε δύο βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Πρώτον, η αξιολόγηση του κανονισμού εκ των υστέρων. Θα προσέξουμε ιδιαίτερως ε, συνέπειες που δεν είχαμε ε, θελήσει ή κενά ε, στη νομοθεσία του Solvency 2, ειδικώ αν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον καταναλωτή, η κερδοφορία, το κατά πόσο ταιριάζει το προϊόν στον καταναλωτή. Όλα αυτά θα τύχουν της προσοχής μας. Και δεύτερον, σύγκληση των εποπτικών πρακτικών. Παρόλο που σημειώσαμε πολύ σημαντική προόδο, για τη δημιουργία μιας κοινή ευρωπαϊκής εποπτικής κουλτούρας παραμένουν εμπόδια στο δρόμο μας, ωστόσο τα ωφέλη της σύγκλησης είναι ξεκάθαρα. Ε, η δουλειά μας έχει αρχίσει και αποδίδει, διότι ενισχύει την ποιότητα και τη συνέπεια της εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια εσωτερική ενιαία αγορά. Η ποιότητα της εποπτείας δεν είναι τοπικό ζήτημα μόνο, αλλά και ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό σύστημα επόπτευσης είναι τόσο ισχυρό όσο ισχυρός ή αδύναμος μπορεί να είναι ο πιο αδύναμος του κρίκος. Και η αξιόπιστη και ανεξάρτητη εποπτεία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών, άρα είναι απαραίτητο και προς το συμφέρον όλων να έχουμε τους επαρκείς πόρους έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι εθνικές αρχές κάνουν σωστή εποπτεία με βάση το κίνδυνο. Τα επόμενα χρόνια ε, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το ότι στηρίζεται το έργο μας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Εργασιακών Συντάξεων. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε και στο μέλλον σε θέση να συμβάλλουμε στη συζήτηση με εσά προς όφελος της σταθερότητα και της προστασίας του καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ, Γκάμπριελ, για την πολύ ενδιαφέρουσά σα παρέμβαση. Και Περιμένουμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ε, ε, στα θέματα που θίξατε. Να πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Να διευκρινίσω ότι πρώτα θα είναι δύο, λεπτά και μετά θα είναι τρία. Άρα θα κλείνω το μικρόφωνο στα δύο λεπτά. Ο καθένας έχει δύο λεπτά να διατυπώσει την ε, ερώτησή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μείνω κάτω από τα δύο λεπτά. Να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές. Όμως λόγω των περιορισμών του χρόνου θα απευθύνω μια ερώτηση στον Γκάμπριελ Μπερναρντίνο. Καθώς ήμουν τότε εισηγητής για την οδηγία Omnibus 2. Η οποία από 1η Πρώτου 2016 θα πρέπει να εφαρμοστεί. Πλέον δεν ε, υπάρχουν άλλα περιθώρια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον πρόεδρο της ε, ε, ΕΙΟΠΑ κατά την άποψή του πώς βλέπει το ότι η Κομισιόν ε, ζήτησε να παραβιαστούν κάποιες ε, προθεσμίες για την εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών. Η Κομισιόν υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και ε, όπως και όλες οι υποτικές αρχές δεν επιτρέπεται να παραβιάζει το υφιστάμενο δίκαιο. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς βλέπετε την αλλαγή που έχει ανακοινωθεί στην πράξη κατεξιοδότηση. Ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και όπως ξέρετε ένα από τα βασικά πράγματα από την ε, δική μας ε, την πλευρά και νομίζω πως το είχαμε πει ξεκάθαρα και το λέω πάντα είναι η σταθερότητα των ρυθμιστικών απαιτήσεων αυτή τη στιγμή οπότε οπωσδήποτε εμείς δεν συμβουλεύουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε αλλαγές στις ρυθμιστικές απαιτήσεις που υπάρχουν. Όπως ξέρετε υπάρχουν κάποιοι τομείς που προέρχονται και από την ε, Ένωση Κεφαλαγορών ε, και υπήρχε ένα θέμα που αφορούσε νομίζω αν δεν κάνω λάθος το μεταβατικό μετοχικό κεφάλαιο και εξετάζονταν κάποιες αλλαγές στο επίπεδο 2 ενημερώσαμε και το Κοινοβούλιο και ακριβώς για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να αποφύγουμε την σύγχυση αυτή γιατί δημοσιεύουμε κάτι και μετά έρχεται η Κομισιόν με κάτι διαφορετικό που θα πρέπει να ενσωματωθεί μετά στο ITS. Οπότε είμαστε σε συνεργασία και με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο και αν γίνουν αλλαγές της κατά κατεξιοδότηση θα σας αναφέρουμε οπωσδήποτε τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω πως ε, θα είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τη γενικότερη πολιτική της σταθερότητας. Και μετά αφού εφαρμοστεί το νέο καθεστώς ε, προβλέπεται σε αυτό μια περίοδος αναθεώρησης ακριβώς για να παρακολουθούμε τις συνέπειες που θα έχει η οδηγία για την εφεργειότητα 2. Μπορκάτ, ναι. ναι. Υπάρχει λίγος χρόνος, θα ήθελα να απαντήσω εγώ θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα η ΕΙΟΠΑ να μας ενημερώνει και να μας είχε ενημερώσει απευθείας εδώ στο Κοινοβουλίο. Και θα ήθελα να παρατηρήσω πως στην περίπτωση που αναβληθεί η εφαρμογή των ε, τεχνικών προδιαγραφών ε, λόγω αλλαγής της πράξης καθεξιοδότηση θεωρώ πως βρισκόμαστε σε νομική γκρίζα ζώνη, να μην πω παραβίαση των ε, αποφασισμένων και να προσθέσω και κάτι άλλο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το Κοινοβούλιο χρειάζεται τουλάχιστον τρεις μήνες χρόνο για την εξέταση των πράξεων κατεξιοδότηση. Πρέπει και αυτό να το υπενθυμίζω, νομίζω. Right. Perfect. Um, now next speaker, Elisa Ferreira. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα του τρει εκπροσώπου εδώ και τη δουλειά που έχουν κάνει σε αυτά τα χρόνια ε, ξεκινήματος μιας νέας ε, λειτουργία. και έχω κάποιες ερωτήσεις, ε, είτε θα μου απαντήσει το καθένα ξεχωριστά, πάντως απευθύνονται σε όλους. Τώρα, περιορισμοί γνωστοί του προϋπολογισμού σε σχέση με την εκτέλεση των των καθηκόντων που σας ζητούνται. Είναι εντάξει μετάφραση, μάλιστα. Ε, έχοντας αυτό υπόψη ποια είναι η δική σας στρατηγική και ποια νομοθεσία επίπεδου 1 μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αφαιθεί ή να παραβλεφθεί λόγω της έλλειψης πόρων. Δεύτερον, στην κοινοβούλιο, στην έκθεση που συνέταξε ο συνάδελφος Γκικούλ, του προτείνει να ενισχυθεί η εντολή των ΕΖΑΣ ε, ενισχύοντας και τις δυνατότητές τους να προβαίνουν σε διαμεσολάβηση υποχρεωτική ή μη και άρα να έχουν περισσότερες εξουσίες. Μέχρι ποιο βαθμό είναι κάτι τέτοιο βιώσιμο και εφικτό και ποιοι είναι οι όροι για να συμβεί κάτι τέτοιο. Τρίτον, όλοι σας μιλήσατε για την ανάγκη να υπάρχει μια εναρμόνιση των πρακτικών εποπτείας ε, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι προφανές, αλλά σε ποιο βαθμό τα τρία αυτά σώματα έχουν δημιουργήσει θέση, ε, μεθόδους εργασίας έτσι ώστε σε ένα θεσμικό όργανο το οποίο λειτουργεί μέσα σε, όπως τα δικά σας να μπορέσει να επιτύχει αυτό το στόχο. Να μπορέσει δηλαδή να, έχει μια, να έχετε μαζί μια συντονισμένη θέση γιατί αυτό είναι στην ουσία ένα πολύ κεντρικό ζήτημα έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή στρατηγική στην εσωτερική αγορά για τα μεγάλα θέματα και τις μεγάλες ε, συστημικές εταιρείες. Σας ευχαριστώ. Να σας να απαντήσω πρώτα στην πρώτη σας παρατήρηση για τον προϋπολογισμό και την διαμεσολάβηση. Ε, για το προϋπολογισμό και γι' αυτό υπήρχε, ήταν, αυτός ήταν ο λόγος και για την κοινή διατύπωση στις ε, δηλώσεις της κοινή Επιτροπής όσον αφορά τις ανησυχίες μας ε, για τα τρέχοντα ε, επίπεδα του προπολογισμού. Με αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε εμείς να υλοποιήσουμε, τα, να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας. Όπως και ο Ανδρέα, όπως και ο Γκάμπριελ, από νωρίς έχουμε δηλώσει ποιε είναι οι νομικέ απαιτήσει, τι οποίε δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αν δείτε την προηγούμενη, τη δήλωσή μα για την προηγούμενη χρονιά, ήδη υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα επιτύχουμε το 2015 και παρομοίω θα συμβεί και για το 2016. πιο, το πιο λογικό για να καθυστερήσει είναι ε, εκείνα που, εκείνα που απορροφούν ιδιαίτερα πολλούς πόρους και έχουν να κάνουν με την ε, ε, τεχνολογία της πληροφορίας, τη συλλογή στοιχείων. Υπάρχουν όμως απαιτήσει για συλλογή στοιχείων που είναι επιτακτικές και απορροφούν πόρους IT ε, και αν δείτε από τον προπολογισμό μας για φέτος υπάρχει ένας κατάλογος δραστηριοτήτων που έχουμε αναβάλει. Όμως ο όγκος εργασίας που αναβάλλεται αυξάνεται. Ε, ελπίζαμε ότι του χρόνου θα μπορούσαμε κάπως να καλύψουμε αυτές τις νομικές απαιτήσεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται με τον προϋπολογισμό για το 2006 θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να καλύψουμε πράγματα τα οποία είχαμε συμφωνήσει ότι θα υλοποιηθούν το 2015. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα καθήκοντα και ο προπολογισμό δεν είναι ευθυγραμμισμένα και δική μα προτίμηση θα ήταν να εξασφαλίζεται ότι ο προπολογισμό συμφωνεί με τι απαιτήσει στι νομικέ μα εντολέ. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάποιες από τη... κάποια από τα καθήκοντά μα δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν. Για το τμήμα της διαμεσολάβησης αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ε, και πρέπει να είμαι ειλικρινή μαζί σας, δεν έχουμε προχωρήσει σε επίσημη κατάσταση διαμεσολάβησης, αλλά ατύπω το έχουμε κάνει αυτό. Ε, εάν κάτι τέτοιο τυποποιηθεί, μάλλον θα ήταν αρνητικό. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει λοιπόν ρητά ως μηχανισμό, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις άτυπης διαμεσολάβησης που ήταν πολύ παραγωγικές και χρήσιμες. Σας ευχαριστώ. Σύντομα, αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Αντρέα, ναι, πολύ σύντομα για το θέμα του προϋπολογισμού. Είμαστε στην ίδια γραμμή, όπως και ο συνάδελφος στην, ε, της ΕΣΜΑ. Στη δική μας περίπτωση όμως υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα, ότι δηλαδή με την ε, δυνατότητα της μεταγραφής των, της προσωπικής συμβολής ε, πραγματικά βουλιάζουμε. αν ε, δεν υπάρξει σημαντική αλλαγή στον προπολογισμό μας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς θα λειτουργήσουμε του χρόνου που είναι κρίμα γιατί πραγματικά θέλουμε να κλείσουμε τα βιβλία για την οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομεριών της ε, αναδιάρθρωσης. Πιεζόμαστε και από τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να κλείσει αυτή η υπόθεση για τη διαμεσολάβηση ε, διάβασα την έκθεση του Σπεν του για την διαμεσολάβηση υπήρξαν κάποιες τέτοιες υποθέσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν φτάσαμε σε ψηφοφορία επειδή η δεσμευτική φύση ήταν εκεί δεσμευτικό αποτέλεσμα δηλαδή ήταν τότε, ήταν πολύ σημαντικό οι αρχές να φτάσουν σε συμφωνία, να συμφιλιώσουν, να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους πριν να χρειαστεί να φτάσουν σε ψηφοφορία. Το γεγονός ότι η EBA είχε τη δυνατότητα να θέσει κάτι σε ψηφοφορία ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα, για τη σύγκληση των σωμάτων καθώς προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Φυσικά η Τραπεζική Ένωση είναι μεγάλη αλλαγή και προσπαθούμε ακριβώς να καταλάβουμε πού μπορούμε εμείς κάτι να προσθέσουμε. Και θα έλεγα δύο τομείς είναι αυτοί που ελκύουν την προσοχή μας. Η μία είναι η κατάρτιση όπου αναπτύσσουμε κοινή πρωτοβουλία με το ε, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Πολύ το τονίζουμε αυτό. Και το δεύτερο είναι η σύγκριση των επιδόσεων το έχουμε κάνει αυτό. Το να δίνουμε δηλαδή συγκεκριμένες ε, στόχους ε, να δουν που έχουν φτάσει είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την σύγκληση. Ευχαριστώ. Και ο Γκάμπριελ. Ναι, για τα όσα υπόθηκαν και βέβαια για το προπολογισμό, ήδη το είδαμε από το 2015 ποιε είναι οι συνέπειε στην εφαρμογή του Solvency 2, όπου αρκετά πράγματα χρειάστηκε να τα αφήσουμε. Όπω α πούμε η ανάπτυξη τη πλατφόρμα IT, που είναι πολύ σημαντική για τη συλλογή των πληροφοριών και να μπορούμε να κάνουμε τη σωστή ανάλυση κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εκεί έπρεπε να καταργήσουμε διάφορα βήματα και για την κατάρτιση των εποπτών, που είναι επίση πολύ σημαντικό ζήτημα για την εφαρμογή του Solvency 2 και ούτω καθεξής. Προχωρήσαμε και φτιάξαμε αυτή την έκθεση που σα στείλαμε, που προερχόταν από την Omnibus 2, και είδαμε ότι, για το, εκεί μάλλον λέγαμε ότι για το 2016 και αργότερα θα έχουμε προβλήματα αν δεν έχουμε τους κατάλληλους ε, πόρους για να κάνουμε τις ε, σταθμίσεις, ε, ε, την αξιολόγηση των εγγυήσεων, όλα αυτά, όλες οι αναλύσεις, όλα αυτά θα αμφισβητηθούν. Είναι ένα διορθωτικό στοιχείο το οποίο έχουμε συζητήσει επανελειμμένως. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου, το στοιχείο της υποπτικής σύγκληση, τουλάχιστον για τις ασφαλιστικές, είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είμαστε μόνο στον τραπεζικό τομέα που έχουμε την SSM. Ε, η σύγκληση των υποπτικών αρχών ούτως ή άλλως για τις ασφαλιστικές θα έρθει σε εμά. Και έχω τώρα τέσσερις ανθρώπους στην ομάδα εποπτείας. Έχω τέσσερις έμπειρους επόπτες. Πώς μπορώ να κάνω σύγκληση των εποπτικών αρχών με τέσσερα όλα και όλα άτομα. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους με την εμπειρία αυτή και ιδιαίτερα όσον αφορά την εποπτεία των εσωτερικών προτύπων, γιατί η παρακολούθηση αυτών θα είναι πολύ σημαντική, γιατί εκεί τίθεται τα θέματα ισοτιμίας, ισότιμου πεδίου. Το ίδιο που, θα, που, το είδαμε στις στον τραπεζικό τομέα θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις ασφαλιστικές και τέλος για την διάθεση της κοινή επιτροπής. Ελπίζω ότι το 2016, αν είμαι εκεί, ε, αν είμαι σε αυτή την κοινή επιτροπή, επιτροπή, ελπίζω πως θα μπορέσουμε α, να συνεργαστούμε στην μεικτή επιτροπή, ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σφίμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προετοιμαζόμενοι για αυτή την ακρόαση ως πολιτική ομάδα αντιληφθήκαμε ότι έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για τους προέδρους και πρέπει να περιοριστούμε στα πέντε λεπτά μόνο. Επομένως μετά θα σας στείλω και γραπτές ερωτήσεις αγαπητοί πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Τα δεδομένα είναι στοιχείο κλειδί για την πληροφόρηση και τα τελευταία χρόνια. Και ε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει βελτιωθεί για το reporting των χρηματοπιστωτικών συνελλαγών. Όσο πιο πολλά δεδομένα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές, τόσο πιο εύκολα θα παρακολουθούν το συστημικό κίνδυνο. Επομένως, από τα 85 παιδεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν πόσα είναι τα ίδια με τα 81 παιδεία που απαιτεί η ΜΥΦΙΡ και πόσα είναι τα ίδια με ναι, αυτά τα πεδία που απαιτεί η MIFID και ε, πόσα τελικά είναι ίδια με τα CSTCs. Εν πάση συμφωνείτε με την αρχή της απλούστευσης και του, της τυποποίησης των σετ δεδομένων. Δεσμεύεστε ότι θα ασκήσετε εξουσία για να ε, ανεβάσετε τα εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα σε αυτά των ε, προτύπων για τα data, για τα δεδομένα. Θα δεσμεύεστε ότι θα υπάρχει όσο το μεγαλύτερη συνέπεια και όλες οι αρχές και οι τρεις αρχές έχουν, ε, δημοσιεύσει, έχουν δημοσιεύσει έγγραφα Q&A, ερωτήσεων και απαντήσεων. Και ε, διαβουλεύονται οι αρχές το RTS και το ITS τις, ε, τους κανονιστικούς, τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα και τα εφαρμοστικά τεχνικά πρότυπα και υπάρχει διαβούλευση και με το Κοινοβούλιο. Όμως το Συμβούλιο των Εποπτών και η κοινή γνώμη μπορούν να συμβουλευθούν ε, τις ερωταποκρίσεις. Μπορείτε να τα εκδώσετε. Ευχαριστώ. Απάντηση θα απαντήσω για το, στην πρώτη σας ερώτηση για τα δεδομένα. Προφανώς, συμφωνώ απολύτως Η αξία της τυποποίησης των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Να τονίσω καταρχάς ότι πράγματι τα αξιοποιούμε. Οι αποφάσεις για την κεντρική εκαθάριση ελήφθηκαν και κάναμε πρόταση για την κεντρική εκαθάριση των παραγωγών και αυτές οι προτάσεις προκύπτουν από τα σετ δεδομένων που μας έρχονται από τα αποθετήρια των τίτλων. Και θέλω να επιβεβαιώσω ότι ήδη ε, τα αξιοποιούμε ιδιαίτερως και τα ε, αξιοποιούν οι θύνοντες που χαράσουν την πολιτική για να συμμορφούνται με τις απαιτήσει για την κεντρική εκαθάριση των συναλλαγών. Με βάση τις εμπειρίες που είχαμε, ήδη σκεφτόμαστε το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη μορφή υπό την οποία παρουσιάζονται, το χρονοδιάγραμμά τους, το πότε εμφανίζονται και πόσο, πόσο είναι να υπάρχει ω δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια με τους ομολόγους. Γιατί υπάρχει μια ομοιόμορφη χρήση παντού. Και δεύτερον, έχουμε μια τυποποιημένη προσέγγιση. Προσπαθούμε ε, εκεί να φτάσουμε. Ε, στοιχεία δεδομένα αναφοράς για χρηματοπιστωτικά εργαλεία και αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς ρευστότητας και για σκοπούς διαφάνειας και όλα αυτά είναι εθνικά προπετούμενα. Το Συμβούλιο όμως συνειδητοποιήσει ότι ε, σε αυτό το πεδίο πρέπει να πάμε σε κοινέ λύσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά επίγον σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε τώρα. Σχεδόν όλες οι αρχές, οι 30, έχουν συμφωνήσει ότι η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η ΕΣΜΑ, θα φτιάξει το λογισμικό θα διαμορφώσει τα τεχνικά πρότυπα δηλαδή για να συμμορφωθούν όλοι με τα προαπαιτούμενα. Επομένω, η τυποποίηση θα είναι ε, ε, πολύ σημαντική στον τομέα αυτό. Ο Ανδρέα, ναι, σας ευχαριστώ για το ερώτημα, για τις ερωταποκρίσεις Q&A. Ε, πολύ συχνά αυτό το παραμελούμε και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στο παρελθόν εκδίδοντο κανόνες και μετά οι τράπεζες τους ε, ε, εφάρμοζαν, καλούσαν μετά τις ρυθμιστικές αρχές της εθνικές και ζητούσαν ερμηνείες. Και οι, ε, ε οι ρυθμιστικές αρχές έθνη καθεμία τη δικιά της ερμηνεία και υπήρχε θέμα συνέπειας. Επομένως, κάναμε μια διπλή διαδικασία ως προς την ερμηνεία, ερμηνεία του πρωτογενούς δικαίου έρχεται η Επιτροπή να παίξει στο παιχνίδι και συμβάλλει στην ερμηνεία της πρωτογενούς νομοθεσίας, ενώ εάν πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες έχουμε ένα δίκτυο γνωμόνων και ειδικών από τις εθνικές αρχές που ασχολούνται με αυτά τα ερωτήματα, τα οποία μετά πάνε στην Τεχνική Επιτροπή και αν υπάρχουν διαφωνίες πάνε σε επίπεδο συμβουλίου και εκεί πλέον αν παραμένουν οι διαφωνίες υπάρχει ψηφοφορία. Μία ευρεία διαδικασία που εμπλέκει όλες τις αρμόδιες αρχές και ο κλάδος ξέρετε στην αρχή ήταν επιφυλακτικός γιατί θεωρούσε ότι αυτό ε, κάνει τη διαδικασία λήψης τεχνικών απαντήσεων πολύ πιο χρονοβόρα. Όμως έλαβα μία επιστολή από τρεις τραπεζικές ενώσεις οι οποίες με συνεχάρηκαν για το γεγονό ότι μπορέσαμε να δώσουμε γρήγορα απαντήσεις και μάλιστα ομοιόμορφες για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το εισπράττουν ως πρόοδο και από την δική τους πλευρά. Ο πρόεδρος της ΕΙΟΠΑ, η διαδικασία μας είναι παρόμοια με αυτό το οποίο περιέγραψε ο Ανδρέας και πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο η συνέπεια και αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε την οδηγία για 2 και έχουμε διάφορες ερωτήσεις από τους ανθρώπους του κλάδου που αντιμετωπίζουν την ΕΙΟΠΑ όπως ανέφερε ο Ανδρέας και βεβαίως αυτή είναι μια ερμηνεία ίσως που είναι θεμελιώδης. Τώρα για την τυποποίηση και τα δεδομένα και να μην κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά να αναφέρω ένα απλό πράγμα για τις απαιτήσει αναφοράς από πλευρά της φερεγγιότητας 2. Τρία χρόνια εργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι ώστε οι νέε στατιστικέ απαιτήσει για τι ασφαλιστικέ εταιρείε να είναι ευθυγραμμισμένε. Και τελικά αυτό αποδείχθηκε πω ήταν φανταστικό από πλευρά αποτελεσματικότητα γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ουσιαστικά τώρα έχει λάβει τα ίδια στοιχεία από τα οποία ζητούσαμε από τον κλάδο. Οπότε δεν γίνονται δύο φορέ ε, τα ίδια πράγματα και αυτό που σα ανέφερα έχει παίξει τεράστιο ρόλο. Σα ευχαριστώ κυρία Σελβιγκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους ε, που ήρθατε και θα είμαι σύντομη. Κύριε Ενγριά, αν έχετε πρόβλημα με την ισοτιμία, με την αλλαγή του ευρώ, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό. Η πλειονότητα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου είχε ψηφίσει η έδρα ε, των τριών εποπτικών αρχών να είναι στη Φραγκφούρτη. Μπορούμε όμως να επανέλθουμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Σβέν Κίγκολντ, η Μάντι και άλλοι θα, θα συντάξουν μια έκθεση από κοινού για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνούς, διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τι πιστεύετε, έχετε τα κατάλληλα εφόδια, τι μπορείτε να μας πείτε. Σταματώ και μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γραπτός και μόλις υπάρξει έκθεση θα σας τη στείλω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω για την έδρα τι να σας πω, εκτός αν θέλετε να μετακομίσουμε στην ε, Φραγκφούρτη. Λοιπόν, ποιος θα είναι να απαντήσει τώρα, Στίβεν. Ευχαριστώ για το ζήτημα των ε, πόρων τώρα για το διεθνές ε, κομμάτι. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το που αφιερώνουμε τους πόρους μας σε διεθνείς δραστηριότητες. Το κάνουμε πάρα πολύ στοχευμένα, όπως φαντάζεστε εστιάζουμε παραδείγματο χάρη σε ύψο αξιολόγηση, ε, παράγωγα, ε, εκεί πέρα κυρίω ε, καταβάλουμε προσπάθειες ακριβώς γιατί θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί με το που ξοδεύουμε τους πόρους μας. Ένα άλλο στοιχείο για τον διεθνή συντονισμό είναι ο συντονισμό και διάλογος και μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και κρατών διεθνώς και αυτό σχετίζεται με το ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, όταν υπάρχει ε, εποπτική ή νομοθετική δουλειά που πρέπει να γίνει να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα οποία υπάρχουν ήδη από διεθνείς οργανισμούς. Ευχαριστώ Ανδρέα. Εγώ ευχαριστώ ε, να συνεισφέρω στην έκθεση την οποία γράφεται. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι πως ε, τα ζητήματα των πόρων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το θέμα της ισοδυναμίας που έχει σημασία γιατί αν ε, δεν το κάνουμε αυτό για κάποιες ε, περιοχές οι τράπεζες οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε αυτές τις περιοχές θα έχουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και έχουμε δυσκολίες στο να βρούμε προσωπικό και απευθυνόμαστε και σε εθνικές αρχές Και εκεί πέρα ναι, έχουμε δυσκολίες. Να πω λοιπόν πως είμαι ικανοποιημένος γιατί σε κάποιους ε, τομείς που έχουμε κάνει ε, ευρωπαϊκή δουλειά, π.χ. στο θέμα της ε, τιτλοποίησης ή τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγηση κινδύνου, καταλήξαμε σε μια ευρωπαϊκή θέση η οποία ήταν ενιαία σε παγκόσμιες διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος από τον ρόλο μας ε, στις ε, διεθνείς επιτροπές. Νομίζω πως μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι για την ε, διεθνή συνεργασία. Έχω κάποια καλά και κάποια άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι πως από την αρχή το 2011 υπήρχε μια συμφωνία στο Υποπτικό Συμβούλιο πως ο πρόεδρος θα έπρεπε να έχει κάποια θέση στον διεθνή διάλογο. Οπότε μπορούμε έτσι να συνεισφέρουμε σε μια κοινή βάση ευρωπαϊκών θέσεων και αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάπτυξη των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις ασφάλειες διεθνώς. Βεβαίω το πρόβλημα είναι πως έχουμε περιορισμένη παρουσία λόγω έλλειψης πόρων. Έχουμε πάνω από 20 τομείς εργασίας και παρακολουθούμε κυρίως τις, τους δύο. Και το άλλο θέμα είναι ο ρόλος βεβαίως του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας γιατί αποκτά ένα σημαντικό ρόλο και στην πλευρά των ασφαλιών κοιτάνε κάποια ζητήματα όπως ε, η άσωση των τραπεζών έχουμε απευθύνει κάποια ερωτήματα στην Κομισιόν και νομίζω πως στο μέλλον Σιλβί ε, θα είναι σημαντικό αυτό το θέμα για την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκολτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Πάντα με χαρά σας ε, υποδεχόμαστε εδώ. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Όταν κοιτάμε το τι έχουμε επιτύχει στους ε, τομείς ε, της πιο έντονης και συνεκτικής εποπτείας, ο κίνδυνος είναι μήπως παγκόσμια προφίλ παρόμοια με συγχωρείτε προφίλ κινδύνου αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους κλάδους. Είτε μιλάμε για το κεφάλαιο, την ρευστότητα και τις εποπτικές ε, πρακτικές. Στην πράσινη βίβλο για την σκιώδη τραπεζική ετέθη το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω συγκεκριμένα μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και τραπεζών ε, μήπως οι ασφάλειες πηγαίνουν στην δουλειά των ε, των τραπεζών λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Και αναρωτιέμαι αν έχετε σκεφτεί να εργαστείτε συστηματικά στις ε, ρυθμιστικές και εποπτικές διαφορές μεταξύ των κλάδων. Κατόπιν, Στίβεν, με συγχωρείς, αλλά το καλοκαίρι έλαβα άλλο ένα έγγραφο από ένα λόμπι το οποίο δεν θα είχε δικαίωμα να λάβει το Κοινοβούλιο. Οπότε ενισχώ ότι οι λομπίστες έχουν εσωτερική πρόσβαση στις υπηρεσίες που δεν έχει το Κοινοβούλιο. Και δεν έχουν και άλλα λόμπι. Μήπω μπορούν να δεσμευτούν οι τρεις αρχές ότι θα έχουν μια σαφή, ξεκάθαρη κοινή πολιτική για το τι θα κάνουν με τους ενδιαφερόμενους ε, τους εξωτερικούς όμως. Και να είστε επίσης σαφείς ε, με ποια λόμπι συνεργάζεστε και να ξεκαθαρίσετε πως ε, δεν θα κανονίζονται συναντήσεις με άτομα τα οποία δεν θα είναι εγγεγραμμένα στο ε, μητρό λόμπι. Ναι, ίσως Ευχαριστώ Ζέν, για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως είπαμε πράγματι το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και αναζητήσεις απόδοσης είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι πρώτη μας προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Και καθορίσαμε και ένα πλαίσιο για τη μακροπροληπτική αντιμετώπιση και του ασφαλιστικού τομέα στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Συστημικής Σταθερότητας. Υπάρχουν τρεις στόχοι λοιπόν. Πρώτον, βεβαίως, θεωρούν πως χρειάζεται μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του κλάδου και εδώ πέρα παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Δεύτερον, να μειωθεί ο κίνδυνος από την αναζήτηση αποδόσεων και τρίτον, να μην ενισχύσουμε τις κυκλικές τάσεις. Και βεβαίως όταν συζητούσαμε και τον κανονισμό Omnibus 2, το ζήτημα αυτών των παραγόντων που ανέφερα, δηλαδή το να η ανθεκτικότητα και να μην έχουμε κύκλικες ε, ε, κινήσεις είναι δύο πράγματα αντιφατικά. Οπότε υπάρχει το ζήτημα της ε, οδηγίας 2, αλλά κάνουμε περισσότερα πράγματα στο πλαίσιο των τεστ κουπόσεων, των λεγόμενων stress test. Στο πλαίσιο τώρα των διασυνοριακών και διατομιακών κανονισμών. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο οπωσδήποτε και θα συνεχίσουμε να το προσέχουμε ειδικά όσον αφορά τις μικρορυθμίσεις που κάνουμε ειδικά στην περίπτωση στην οποία μπορεί κανείς να επιλέγει ρυθμιστικό περιβάλλον αλλά να σας πω κάτι δεν είναι ίση στάθμιση όλων των κινδύνων γιατί το πλαίσιο διαφέρει Παραδείγματο χάρη, η φερεγγιότητα 2 βασίζεται στην ε, αποτίμηση της αγοράς όλων των στοιχείων που υπάρχουν σε ένα χαρτοφυλάκιο, κάτι το οποίο δεν ισχύει στον τομέα των τραπεζών. Όπως είπατε όμως, ε, αυτό είναι κομμάτι της αναθεώρησης της φερεγγιότητας 2 και μάλιστα αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε ταυτόχρονα στον τομέα της ε, τιτλοποίησης έτσι ώστε οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ε, το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένες. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ στην διαρροή που, ανε, που ανέφερε ο Σβέν. Εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, διαρροές γιατί όπως είπατε δεν έχουμε μετά ίσως όρους ανταγωνισμού αν υπάρχει η δυνατότητα ε, να συνεισφέρουν ε, οι ενδιαφερόμενοι, αυτό πρέπει να ισχύει για όλους και όχι για κάποιους λίγους. Ε, θα πρέπει να τονίσω πως τα έγγραφα αυτά δεν είχαν συμφωνηθεί από το ΔΣ, ήταν στο επίπεδο του προσωπικού, ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να αποφευθούν αυτές οι διαρροές. Είναι κατά του κανονισμού μας που δεσμεύει βεβαίως όλα τα μέλη του ΔΣ και οπωσδήποτε και το προσωπικό και κρυπτογραφούμε τα έγγραφα και βάζουμε και υδατογράφημα επάνω οπότε η διαρροή αυτή δεν, οπωσδήποτε δεν συμφωνεί με την πολιτική μας και δεν είναι εύκολο αυτό γιατί ε, μπλέκεται το όλο το προσωπικό στην ε, κατάρτιση αυτών των εγγράφων αλλά όπως είπαμε πρέπει να υπάρχουν ίσοι και αν υπάρχει η δυνατότητα αντίδρασης να αντιδρούν όλοι ανοιχτά. Τώρα, για το δεύτερο που αναφέρατε, για τις ε, συναντήσεις με ενδιαφερόμενους ε, και συγκεκριμένα τον κλάδο. Ήδη έχουμε δεσμευτεί από το 2011 όλοι οι πρόεδροι και εκτελεστικοί διευθυντές θα δημοσιεύουν στην σελίδα τους συναντήσεις με τον κλάδο και από όσο γνωρίζω αυτό το τηρούν όλοι. something?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 Κοίταξε, το μόνο που έχω να τονίσω είναι πέρα από τα υπόλοιπα θέματα και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Γκάμπρελ. Στη διάρκεια τη κρίση και πιο πρόσφατα, θα πρέπει να σα πω ότι είχαμε πολλέ ανταλλαγέ πληροφοριών και κάποιε φορέ μάλιστα και συγκέντρωση ε, στοιχείων για τη μετακίνηση εταιριών, όπου ο κανονισμό ήταν πιο σφιχτό στην τραπεζικό τομέα, οπότε πιερνούσαν σε άλλου τομεί. Είναι πολύ αυστηρή λοιπόν η συνεργασία εδώ. Ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ πέρα ο κύριος ε, Μάριο Ντράγκη, ο πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως ε, η κριτική ασκήθηκε κυρίως προς την κατεύθυνση της δημιουργίας χρήματος. Το ερώτημα μου λοιπόν απευθύνεται προς, τους κυρίους, προς τον κύριο Μπερναρντίνο γιατί βλέπουμε διάφορες εκθέσεις που λένε πώς τα προβλήματα σας τα εξαιρετικά ταμεία αυξάνονται και βεβαίως αυτό οφείλεται και στην πολιτική των χαμηλών επιτοκίων και σύμφωνα με την πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό θα οδηγήσει νομίζω τελικά σε χαμηλότερες συντάξεις και πόσες πιθανότητες υπάρχουν να μην μπορούν πλέον τα συνταξιωτικά ταμεία να ανταποκριθούν στις ε, υποχρεώσεις τους. Και τώρα για τον κύριο Ενρία το επόμενο ερώτημα. Η FSMA επίσης εποπτεύει και μεγάλες τράπεζες όπως η BNP Paribas ειδικά όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Θεωρείτε πως θα πρέπει να παρακολουθείτε το τι γίνεται στο Βέλγιο στενότερα ή θεωρείτε πως επαρκεί μέχρι στιγμής δράση της Βελικής Υποπτικής Αρχής. Σας ευχαριστώ. Γκάμπριελ, όπως είπα, βεβαίως το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων είναι από τα βασικά ζητήματα ε, στην ε, ημερήσια μας διάταξη. Επιπλέον βέβαια, επίσης χρειάζεται να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ε, και παράπλευρες επιπτώσεις από τις, μικρο, τις μικροπολιτικές που έχουν σχεδιαστεί και τις νομισματικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί. Βλέπουμε λοιπόν κάποιο κίνδυνο στις τιμές ε, λόγω της ρευστότητας και αυτό χρειάστηκε να το εξετάσουμε, να δούμε δηλαδή τις τιμές των διαφόρων προϊόντων και να δούμε πώς σχετίζονται μακροπρόθεσμα με το μακροπρόθεσμο στοιχείο, αν είμαστε στη διαδικασία δημιουργίας πιθανών φουσκών ή όχι, αυτό το παρακολουθούμε ε, και το αναφέρουμε στις συμβουλές μας όσον αφορά τις εκθέσεις ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τώρα όσον αφορά τις συνέπειες ε, αυτό το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων έχει και μια δομική συνέπεια στα επιχειρηματικά μοντέλα. Γιατί αν δούμε ας πούμε τις ασφαλιστικές εταιρείες ασφάλεια ζωής που προσφέρουν και προσφέρουν πραγματικά μονοκορπρόθεσμες εγγύσεις, αυτές οι εγγύσεις τώρα αμφισβητώνται λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η δυσκολία εδώ είναι να κατανοήσουμε ποια θα είναι η εξέλιξη των ε, επιτοκίων. Και το είπατε σωστά, ε, το είπαμε και το είδαμε και στις δοκιμές αντοχής και προσπαθήσαμε εδώ να συλλέξουμε τα στοιχεία, γιατί εδώ ε, περιέχονται δύο κίνδυνοι. Ο ένας είναι αν αυτή η περίοδος κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια και έχουμε τελικά μια νέα αξιολόγηση του, των πριμ κινδύνου στην αγορά τότε οι ασφαλιστικέ εταιρείε θα βρεθούν σε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό είναι ένα άσχημο σενάριο, να συνεχιστεί δηλαδή επαόριστο αυτή η κατάσταση και άρα η επαναξιολόγηση των, των ασφαλίστρων κινδύνου. Είδαμε, το έχουμε συζητήσει με διάφορες ομάδες, ότι αυτό θα ήταν μια πρόκληση. Το άλλο θέμα είναι όταν θα αυξηθούν τα επιτόκια. Και αν υπάρξει μια ξαφνική κίνηση, τότε πάλι οι ασφαλιστικέ θα έχουν πρόβλημα. Γιατί μια απότομη κίνηση βέβαια θα, καταστήσει, θα, θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των προϊόντων του συζητάμε με την Κεντρική Τράπεζα και έχουμε καταστήσει σαφέ ότι εντάξει κάποια μέρα των ημερών θα αυξηθούν τα επιτόκια αλλά παρακαλούμε αργά αργά, σιγά σιγά γιατί διαφορετικά ε, γιατί κάτι τέτοιο θα έχει νόημα για τη σταθερότητα του τομέα των ασφαλίσεων. Τέλος, για τα θέματα αφαιρεγιότητας και εδώ βεβαίως ε, ε, μπορεί να υπάρχουν συνέπειες για τις εταιρείε που έχουν αντασφαλίσει δεσμεύσεις στο παρελθόν θα έχουν προβλήματα αφαιρεγιότητας γιατί στα τεστ δοκιμή δεν έχουμε δει μόνο τα θέματα αφαιρεγγιότητας και εκεί είχαμε περίπου 14% των εταιριών που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις αφαιρεγγιότητας που θα προκύψουν από τη Solvency 2, αλλά αυτοί προσωπεύουν γύρω στο 3% του συνόλου των, του συστήματος. Φαίνεται να μην είναι δηλαδή πολύ σημαντικό ζήτημα, ωστόσο προσπαθούμε να μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ανδρέα για την ιδιαίτερη παρατήρηση για την απόφαση του Βελγίου. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι σύμμορφο με την ευελιξία που ε, έχει αφαιθεί στις εθνικές αρχές. Ε, όταν δηλαδή υπάρχουν χαμηλά επιτόκια μπορεί όντως να δημιουργηθεί μία φούσκα ε, στην αγορά κινήτων και έτσι δίνεται δυνατότητα στις αρχές να μπορέσουν να τροποποιήσουν τα επιτόκια και γι' αυτό και υπήρξε αυτή η αλλαγή στη βελγική προσέγγιση. Εν γέννη θα έλεγα ότι η ανησυχία μας είναι ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τη ίδια υπερθέρμανση αυτή της αγοράς των ακινήτων σε διάφορες κράτη-μέλη ε, δημιουργείται με διάφορα εργαλεία. Σε κάποια κράτη έχουμε ε, αναλογίες ε, ε, Εισοδήματο με με, επιτόκια, με διάφορους τρόπους εν πάση περιπτώσει επηρεάζεται η αγορά. Ο Κούναρ Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήματα να θέσω στον κύριο Ενρία. Καταρχάς, ποια είναι η απόψή σα για την εισαγωγή του ΤΙΛΑΚ σε σχέση με τη συζήτηση για τον ορισμό του MRL και σε σχέση με το BRG, τη Total Loss Absorbing Capacity. Και ως προς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από πλευράς εποπτικής αρχής, τι λύπη πιστεύετε στα, στους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουμε. Και ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της εποπτείας. Ε, ποιο πρόβλημα έχουν οι κανόνες ή ο τεράστιος όγκος αν θέλετε αυτών και δυσχεραίνουν την εποπτεία. Κοιτάξτε το TILAC σε σχέση με το MREL είναι προαπαιτούμενο για συστημικές τράπεζες υποχρεωτικό παγκοσμίω. Εμείς αξιολογούμε τα MREL έτσι όπως είναι στο BRDD, στην οδηγία της σχετική για ε, ανάκαμψη και εξυγίαση περισσοτικών ιδρυμάτων. θα πρέπει το MRL δηλαδή οι αρχές να το προσαρμόσουν στην ε, κατάσταση της κάθε τράπεζας. Για συστημικό σημαντικές τράπεζες ίσως υπάρξουν προαπαιτούμενα που θα ταυτίζονται με το TILAC που είναι τα ε, προαπαιτούμενα παγκοσμίω. Εγώ προτιμώ δηλαδή την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τα MRL και όχι τόσο το TILAC γιατί η οδηγία αυτή είχε να κάνει με την διάσωση και εξυγίαση ε, των τραπεζών, ενώ το θύλακ είναι ένα πιο, μια πιο αφηρημένη έννοια. Βεβαίως και, και οι δύο έννοιες μπορούν να συνάδουν και μπορεί ε, να χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή διακρατήσει τίλακ μεταξύ τραπεζών, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε με τα δικά μας πρότυπα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει απόφαση. Το δεύτερο σας ερώτημα είναι επίσης δύσκολο, διότι Θέλω προς το παρόν να είμαι ταπεινός. Κατά τη γνώμη μου η μεγάλη προτεραιότητα είναι τα εσωτερικά μοντέλα, να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των χωρών, δηλαδή των εσωτερικών μοντέλων. Οι αναλυτές και οι επενδυτές ανησυχούν, διότι βλέπουν τράπεζες που θεωρούν ότι έχουν ενιαία χαρτοφυλάκια από τη μία, αλλά μετά έχουν διαφορετικά ε, στοιχεία, όπου ε, προκύπτουν διαφορετικά στοιχεία και δεδομένα για αυτές από πλευράς ρευστότητας και άλλων δράσεων. Άρα εκεί υπάρχει κενό στο σύστημα και δεν υπάρχει τόση εμπιστοσύνη. Και ένα μέρος είναι οι εποπτικές πρακτικές και ένα άλλο μέρος είναι οι πρακτικές των τραπεζών και κάνουμε διάλογο με τις τράπεζες και είναι ένας τρόπος η εποπτεία να είναι περισσότερο συνεπής και πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ο, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι το κύριο Ενρία σε σχέση με τις ε, τραπεζικές διαστρωτικές μεταρρυθμίσεις πάνω στις οποίες εργαζόμαστε και πιο συγκεκριμένα το θέμα home host στην αρχική πρόταση για την ε, τραπεζική αναδιάρθρωση πάρα πολλές εξουσίες θα είχε ο ενοποιημένος επόπτης των μεγάλων τραπεζικών ομίλων σε ό,τι αφορά στη λήψη των αποφάσεων για τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών. Τώρα, το Συμβούλιο, αυτό επρόκειτο να γίνει, το Συμβούλιο Ε, υιοθέτησε μια θέση που αποδυναμώνει κάπως την αρχή του ενοποιημένου επόπτη σε ορισμένα πεδία, ε, διότι εκεί πρέπει να γίνει διαιτησία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή από κοινού και ε, σε άλλα πεδία είναι μεγαλύτερη η εξουσία και η αρχή του επόπτη της χώρας άφηξης, το host supervisor. Ποια θα δώσετε τη δυνατότητα στους host επόπτες ανεξάρτητα να λάβουν απόφαση για μέρος των τραπεζικών εργασιών ή μέρος της τράπεζας ε, την οποία φιλοξενούν. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο. Ε, υπό μία έννοια είναι μία, ένα θέμα που προκύπτει ξανά και ξανά κάθε φορά που εξετάζουμε εξετάζουμε τις κοινέ αποφάσεις στο κεφάλαιο, την επάρκεια και την κεφαλαιακή, την επάρκεια ρευστότητα στους διάφορους ομίλους, στις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και το καθεξής. Θεωρώ ότι οι κοινέ αποφάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε προς τα μπροστά σε όλα αυτά τα πεδία. Θα πρέπει ε, οι αρχές να καταλήγουν σε ένα κοινό ψήφισμα, σε μια κοινή απόφαση μάλλον και όσο περισσότερο το νομοθετικό πλαίσιο τους πρόχνει να πάρουν κοινέ αποφάσεις τόσο το καλύτερο. Ξέρετε, ε, στη, κατά διάρκεια της κρίσης είχαμε όλο και περισσότερο υγειονομικούς κλειούς ε, να κλείνουν γύρω από το ένα ή το άλλο πεδίο. Ωστόσο αυτά επιβραδύνουν την πορεία, αν δεν την κάνουν, αν δεν την κάνουν κιόλας κιόλας. Όσο περισσότερο οι αρχές είναι διασφαλισμένες ότι σε περίπτωση κρίσης θα είναι κοινή η προσέγγιση για την αντιμετώπιση ε, των ζητημάτων, τόσο περισσότερο θα είναι έτοιμες οι αρχές αυτές να αποφύγουν μέτρα υγειονομικού κλειού ε, ε, και αποκλεισμού. και... Όσο λοιπόν έχουμε περισσότερο ε, κοινέ αποφάσεις, τόσο λιγότερο θα έχουμε καταστρεπτικά μέτρα όπως ε, είναι αυτά που σας ανέφερα. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι θηκατρικές των ομίλων έχουν πολύ σχετικό αντίκτυπο στις εγχώριες αγορές. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες των αρχών host έχουν συμπεριληφθεί επαρκώς στις ε, αποφάσεις που λαμβάνονται σε συλλογικό επίπεδο. Όσο περισσότερες κοινέ αποφάσεις έχουμε από κοινού αποφάσεις και όσο περισσότερο δεσμευτικές είναι αυτές ε, σε σχέση με την παραδοχή της διαμεσολάβησης ε, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για όλα τα πεδία συμπεριλαμβανομένων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμασούρ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις Προέδρους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Ένα και μόνο είναι το ερώτημά μου, κυρίως στο Στίβεν Μάισμιορ και στην ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Σε ποιο βαθμό οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που επέτρεψαν την υλοποίηση, την εφαρμογή του κανονισμού για το Ταμείο επενδύσεων σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου, σε κοινωνική εταιρική σχέση μεταξύ άλλων έχουν φτάσει σε πιο βαθμό τους αρχικούς τους στόχους και κυρίως στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Αυτά τα εργαλεία είναι κινητοποιήσιμα ήδη ή χρειάζονται κανονιστικό συμπλήρωμα και νομοθετική πρόβλεψη συμπληρωματική για να αξιοποιηθούν. Ευχαριστώ. Ο Στίβεν. Κοιτάξτε, για τον τομέα της ε, διαχείρισης ε, στοιχείων ενεργητικού, οπωσδήποτε θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην συζήτηση για την Ένωση των Κεφαλαίων και την συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και οπωσδήποτε μπορεί να παίξει έναν ρόλο διάβλου χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι αναζητούν κεφάλαια και θα ήθελαν καλή απόδοση για τα κεφάλαια τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία του κλάδου να διαπιστώσουμε πως έχει ήδη παίξει τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν αναπτύσσεται. Κάποιοι το λένε ε, σκιώδη τραπεζική. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο ακριβείς. Θεωρώ πως ε, κάποια στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν ως σκιώδης τραπεζική, αλλά μεγάλα τμήματα του κλάδου συνεισφέρουν στον δανεισμό επιχειρήσεων αν δείτε π.χ. τα διάφορα τμήματα της ε, νομοθεσίας ε, που λέγεται γιουρίκα. Εκεί πέρα περιορίζεται σε κάποιες επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους και θα μπορούσε βέβαια να ε, καλύψει και άλλες μεγαλύτερες. Ένα άλλο σημαντικότερο σημείο είναι να δούμε το τι γίνεται και στα usage και τα FMD, παραδείγματος χάρη όπου απαιτούνται τέλη, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κράτους προέλευσης, αλλά και του κράτους το οποίο δραστηριοποιείται και βέβαια οπωσδήποτε όλα αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αγοραστούν από καταναλωτές λιανικής. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο τους εάν δεν συμμετέχει και ο καταναλωτής, ο τελικός ε, χρήστης. Και βέβαια ε, το να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτού του κλάδου για να έχουν ε, να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες νομίζω θα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για να συνεισφέρουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη. I think, has a lot to do with pensions, so... Ναι, βεβαίω ε, νομίζω πως ε, το θέμα αφορούσε και τις συντάξεις, οπότε θα δώσω τον λόγο στον Γκάμπριελ. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Και νομίζω πως ε, μπορεί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο χρηματοδότηση οικονομίας, να υπάρξουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και βεβαίως να έχουν και αυτοί ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, να μην ε, έχουν τόσο να μην διατρέχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο. Αλλά βεβαίω αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι βιώσιμος. Για να μην χρησιμοποιούμε παραδείγματο χάρη ε, κανόνες ε, και ρυθμιστικούς κανόνες που θα δημιουργούν τελικά ένα κίνητρο το οποίο σε λίγα χρόνια θα μας οδηγήσει σε μια νέα φούσκα και νέα προβλήματα και αδυναμίες. Πρέπει λοιπόν να διδαχτούμε τα λάθη του παρελθόντος. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Συμβουλεύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατηγορία αυτή υποδομών για να μπορέσουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε ένα διώσιμο στοιχείο στο οποίο θα μπορούσαν να κατευθυνθούν και συνταξιδοτικά ταμεία και οπωσδήποτε θα παρακολουθούμε και τα επόμενα χρόνια πώς θα συμβεί όντω αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελίζα Φερέιρα και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τα όσα είπε ο κύριος Ενρία όταν λέει πως ε, η η εποπτεία των τραπεζών ε, έχει οδηγήσει ή μάλλον υπάρχει αίσθηση πως ε, κάποιοι παρακάμπτουν ε, τον κανονισμό μέσω του να μετακινούν τις δραστηριότητε τους σε δομές οι οποίες δεν ρυθμίζονται ή δεν υποπτεύονται. Θεωρείται λοιπόν πως υπάρχει ένα παραθυράκι το οποίο μεγαλώνει όσον αφορά την εποπτεία στην ε, Ευρώπη. Πρώτο ερώτημα προς τον κύριο Ενρία. Αναφέρατε στην ε, παρουσίασή σας μια πάρα πολύ σημαντική ανησυχία, δηλαδή την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστοτικών ιδρυμάτων. και βεβαίω μιλήσετε και για τον ενιαίο μηχανισμό διάσωση τραπεζών. Ποιε είναι οι προοπτικέ λοιπόν. Και αναφέρετε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα όταν λέτε παραδείγματο χάρη η εφαρμογή της αρχής της ε, αναλογικότητα στον τομέα των αμοιβών ε, θέτει ευαίσθητα νομικά ζητήματα τα οποία θα απαιτήσουν αλλαγέ της νομοθεσία Τι ακριβώ εννοείται και προ τον κύριο Μπερναρντίνο το ερώτημά μου σχετίζεται με τα PEPS. Ε ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτό το προϊόν και να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για τις συντάξεις. Σας ε, ευχαριστώ. Λοιπόν, προσπαθήστε να, να απαντήσετε σύντομα γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Καλή τύχη. Μάλιστα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως με το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων ο μη τραπεζικός τομέας αυξάνεται. Αλλά όχι επειδή δεν είναι ρυθμισμένος, απλά επειδή αναζητούν αποδόσεις. Γιατί οι επενδυτές, οι καταθέτες γνωρίζουν πως έχουν πάρα πολύ χαμηλές αποδόσεις από το τραπεζικό σύστημα και προσπαθούν να βρουν υψηλότερες ε, αποδόσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν λέμε πως η ανάπτυξη του μη τραπεζικού συστήματος ε, οφείλεται σε μη ε, ρύθμιση. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, δεν υπάρχει σημαντικός ε, κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος και ίσως υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής εκτίμησης των στοιχείων αυτών, αλλά θεωρώ πως ο κίνδυνος είναι των χαμηλών επιτοκίων, το ότι δεν είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι οι επενδυτές όταν είναι χαμηλά τα επιτόκια. Μάλιστα τα καταφέρατε λοιπόν. Είναι κάπως λίγο πιο δύσκολο για μένα όμως να απαντήσω, λέει ο κύριος Σενρία. Τώρα για την έκθεση όπως είπατε στη σκιώδη τραπεζική. Το ερώτημα για μας είναι κατά πόσον οι τράπεζες ε, επεκτείνονται, επεκτείνουν την έκθεσή τους σε σκιώδες τραπεζικές οντότητες, ειδικά εάν αυξάνεται κάπου ο κίνδυνος. Δεν έχουμε κάπου δεδομένα, οπότε είχαμε ένα έγγραφο διαβούλευσης και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς ε, θα να αποκτήσουμε μια αίσθηση του βαθμού έκθεσης. Οι αντιδράσεις που λάβαμε ήταν έντονες γιατί λέ, μας λένε πως ρίχνουμε άδεια να πιάσουμε γεμάτα και ζητάμε πάρα πολλές πληροφορίες που θα δυσκολεύσουν τις τράπεζες κτλ. Ναι, από τη μία πράγματι προσπαθούμε να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία για να λάβουμε τις πληροφορίες τις οποίες ε, θέλουμε για να δούμε πως μεταφέρεται ο κίνδυνος κάπου αλλού. Τώρα για την εφαρμογή των κανονισμών που αναφέρατε Μπορεί να έγινε ένα λάθος στους ε, αριθμούς. Νομίζω πως ε, ορίστηκαν 24 εθνικές εποπτικές αρχές από 28 κράτη-μέλη και η BRD η οδηγία ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως σε ακόμη περισσότερες χώρες. Νομίζω σε 16 εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Οπότε κατά βάση δεν υπάρχει κάποια διαδικασία για την ε, λύση των τραπεζών και τις μηχανισμούς διάσωση. Οπότε δεν θα γίνει σεβαστή τελικά η προθεσμία του τέλους ε, του έτους. Δεν θέλω να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο της απόφασης. Τώρα για την αναλογικότητα των αμοιβών. Κοιτάξτε, η δική μας η ανάγνωση την οποία έχει επιβεβαιώσει η νομική υπηρεσία της Κομισιόν είναι πως κάποιες διατάξεις οδηγίες για την κεφαλιακή επάρκεια που είχαν αδρανοποιηθεί στο παρελθόν για μικρές τράπεζες ε, ή τα μικρά μπόνους στις κατευθυντήριες γραμμές ε, και στην εθνική νομοθεσία δεν μπορούν πλέον να διατηρηθούν στο εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως η αναστολή των ε, αντιβών ή των πληρωμών σε διάφορα μέσα θα ισχύουν και για τράπεζες οι οποίες δίνουν πόνου λίγων χιλιάδων ευρώ. Θεωρούν πως αυτό ε, είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό και δεν νομίζω πως πραγματικά είναι αυτό το οποίο θέλατε εσείς ε, όταν συντάξατε την οδηγία. Οπότε νομίζω πως το καλύτερο είναι νομίζω να εξαιρέσουμε κάποιες μικρές ε, οντότητες και μικρά μπόνους από τις διατάξεις της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, σύντομα. Οπωσδήποτε εργαζόμαστε σε αυτό το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν που στόχο έχει να υπάρξει μια ενιαία αγορά για αποταμιεύσεις για την ε, συνταξιοδότηση. Δεν έχουμε λύσεις, έχουμε μόνο εθνικές λύσεις και υπάρχουν στοιχεία πως ε, τελικά θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές και θα μειωθεί το κόστος μέσω της ε, ενιαίας αγοράς ως εργαλείο. Και βεβαίως στον τομέα αυτών θεωρούμε πως είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Αυτό βεβαίως μπορεί να συνεισφέρει και σε επενδύσεις πιο μακροπρόθεσμες που οπωσδήποτε χρειάζεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπάρχουν τέτοια προβλήματα βεβαίως Κάνουμε ήδη διαβούλευση. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Είμαστε σε επαφή και με τον κλάδο και με εσάς, κάτι το οποίο μας χαροποιεί και θεωρώ τελικά πως μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να έρθουν σε μεγαλύτερη επαφή με την Ένωση νομίζω πως ε, θα φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και να έχουμε κάτι το θετικό. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, η εμπειρία με τις συντάξεις σε κάποιες χώρες ε, δεν είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ. Γαμπριέλ, πράγματι πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση για αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Ντανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ στη σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να λειτουργήσει το πράγμα και για την ανάπτυξη επίσης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το πλαίσιο, γιατί δεν έχουμε ένα καθεστώ εξηγήσει πέρα από τον τραπεζικό τομέα. Δεν ε, είναι αυτό μόνο πρόκληση για την ΕΣΜΑ, αλλά και για τους υπολείπους. Και μάλιστα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Περναντίνο γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα γίνει με ένα μεγάλο συνταξιδικό ταμείο στοχεύσει σαν από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ή κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και επίσης τώρα εισάγονται αλλαγές στη Solvency 2 και υπάρχουν προτάσεις για την νομοθεσία δεύτερου επίπεδου για την εισαγωγή ενός μηχανισμού phasing in των νέων ε, παραγόντων κινδύνου και όπως μάλλον θα γνωρίζετε οι μη καταγεγραμμένες ε, τα χρεόγραφα θα, είναι πιο δύσκολο, θα καταστήσουν πιο δύσκολο για την κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και προς τον κύριο Ένρια ε, μια ερώτηση που σχετίζεται με το γεγονός ότι τώρα υπάρχει ένας προβληματισμός για ένα νέο είδος περιορισμού της έκθεσης των τραπεζικού τομέα σε θέματα αφαιρικιότητας και των ε, στοιχείων των, των, των κυβερνήσεων έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία ανάλογα με το κράτος μέλος. Να έχουμε δηλαδή διαφορετικά όρια έκθεσης για κάθε κράτος μέλος ανάλογα με την ισχύ τους. Ευχαριστώ. Ε, πολύ καλή ερώτηση που πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Εάν δούμε το είδος πλαισίου από πλευράς τη ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη στιγμή, πραγματικό παραθυράκι που βλέπουμε εμείς εδώ είναι ένα ε, συγκεκριμένο πλαίσιο εξυγίανσης για τις ασφαλιστικές εταιρείε. Δεν σημαίνει που δεν έχουμε κάποια μέσα, αλλά είναι διαφορετικά σε κράτη-μέλη. Έχουμε διάφορες εκπαιδευτικές αρχές, διαφορετικά πλαίσια εξυγίανσης ε, ε, όπως είπατε, το έχουμε αυτό εντοπίσει και το έχουμε αναφέρει στην Επιτροπή πολύ συγκεκριμένα. Μέχρι τώρα κάποιες μικρές εταιρείες έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, αλλά με αυτή την εμπειρία ήδη βλέπουμε ότι θα προκύψουν ζητήματα συνοχής ε, ε, στην εποπτεία και στην ε, αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων. Άλλο θέμα είναι πως δεν υπάρχει καθεστώς ενωτικό για την εγγύηση των ασφαλιστικών πλάνων. Αυτή τη στιγμή εξαρτάται από το κάθε ε, κράτος μέλος. Υπάρχουν ένα σωρό παραθυράκια και διαφορετικές ε, εφαρμογές ε, θα πρέπει δηλαδή να γίνουν ένα σωρό πράγματα ώστε να δεθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο στον ασφαλιστικό τομέα. Για την εφαρμογή του Solvency 2 και την μεταβατική περίοδο που αναφέρατε, αυτό συζητήθηκε εντόνω σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορε μεταβατικέ διατάξει που περιλαμβάνονται στη Solvency 2 ή προς το Omnibus 2. Ξέρω πως υπάρχουν ζητήματα όπως αναφέρατε για παράδειγμα στις μη καταγεγραμμένα στοιχεία ε, βέβαια, ε, εδώ δεν μπορούμε να, εμείς να παρέμβουμε. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε εντόνω, όπως είπα, σε πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, όπως έχω ξαναπεί, εμείς θα μεριμνήσουμε, θα φροντίσουμε ώστε να παρακολουθούμε ε, την κατάσταση και να βλέπουμε αν υπάρχουν συνέπειες και φυσικά θα αναφερόμαστε στο Κοινοβούλιο αν κάτι τέτοιο συμβεί. Ο Ανδρέα, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι δεν αναπτύσσουμε συγκεκριμένα όρια έκθεσης τα οποία να μην είναι σύμμορφα με το γενικό νομοθετικό πλαίσιο και τους κινδύνους που υπάρχουν. Ε, αυτό συνδέεται νομίζω με το θέμα της ευαισθησίας απαιτήσεων για τα κράτη, για παράδειγμα. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Αυτό πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι, πρόσφα... ότι υπάρχει μάλλον κάποιες φορές η παρεξήγηση, η εντύπωση δηλαδή ότι ο κρατικός κίνδυνος δεν καλύπτεται από το ισχύον πλαίσιο. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να πω ότι πολλές τράπεζες που υιοθετούν εσωτερικά μοντέλα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην... Ε, σε αυτούς τους κινδύνους. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν είναι συνεπή. Το είδαμε ας πούμε όταν είχαμε την κρίση κρατικού χρέους, είδαμε ότι δεν ήταν το ίδιο ε, ε, ίδια τη εμείς ε, και στα μελλοντικά μας τεστ αντοχής θα σκοπεύουμε να εισάγουμε ε, εγγύησεις πυλώνα 2 ε, για όταν και εφόσον υπάρχουν ε, κρατικά χρέη. Τώρα, αυτό που δεν καλύπτεται είναι το γεγονός ότι κάποιες τράπεζες έχουν υπερβολική έκθεση στην ίδια τους τη χώρα, στην ίδια, στο, προς το ίδιο τους το κράτος, ας πούμε 5-6 φορές το κεφάλαιό τους. Αυτό είναι ένα θέμα από άποψη, ε, από άποψη πρόληψης. Στην Κομισιόν λοιπόν εξετάζονται αυτά τα θέματα, αλλά δεν θέλω να δώσουν την εντύπωση ότι ενώ αναπτύσσονται τα παγκόσμια στάνταρ, εμεί δεν τα έχουμε καταφέρει. Αλλά πάντω εργαζόμαστε και για αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Διαφοροποίηση ήταν μια καλή πρόταση που υπάρχει. Νομίζω πρέπει να εξερευνηθεί αυτή η λύση. Γιάκοπ Φων Βαϊτσέκερ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, μετά την ερώτηση της Δανούτα Χιούπνερ και εγώ σε αυτό το θέμα θέλω να επανέλθω. Καλώς κατέδειξε το πρόβλημα απουσίας σωστού καθεστώτος για τις ασφαλίσεις όταν υπάρξει πρόβλημα. Ίσως οξυνθούν τα προβλήματα. Και να πω και κάτι παραπάνω. Ενδεχομένως οι ασφαλιστικές εταιρείες κάνουν κάποιες υποσχέσεις, δίνουν κάποιες υποσχέσεις που δεν θα έπρεπε να δίδονται σε βάθος χρόνου. Ορισμένα είδη ε, υποσχέσεων ε, ενισχύσεων ωφελημάτων άνευ όρων και σε βάθος χρόνου δεν θα πρέπει πλέον να διδονται σε βαθος χρονου ορισμενα ειδη υποσχεσεων εύκολα αλλά να είναι εξαρτώμενα από μεγάλες εξελίξεις στο μακροοικονομικό πεδίο. Ε, Ποια είναι η γνώμη σας για τη χρονική πλαισίωση των ασφαλιστικών συμβάσεων που θα συνεχιστεί να επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά. Απάντηση. Πολύ καλή η ερώτησή σας και σας έχω ήδη πει ότι ένα από τα πράγματα τα βασικά που είδαμε από το 2011 και μετά, κάθε φορά που εκδίδαμε γνωμοδοτήσεις και συστάσεις σε σχέση με ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, είναι το θέμα το του διαρθρωτικού στοιχείου, του δομικού στοιχείου στις συμβάσεις και στα συμβόλαια που προτείνει κάποιος οργανισμός. Και στον κλάδο το έχουμε πει επανειλημμένως ότι δηλαδή είναι θεμελιώδες, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εταιρείε να δουν πώς μπορούν να ανακατέψουν την τραπούλα στις επιχειρήσεις τους, στο αντικείμενό τους. Δηλαδή ε, δεν είχαν τιμολογήσει σωστά αυτές τις υποσχέσεις σε βάθος χρόνου και τα options και οι εγγυήσει υπάρχουν, αλλά με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρέπει να υπάρχει η συνέπεια με την αγορά. Όλα αυτά αναδύονται στην επιφάνεια. Αυτό το στοιχείο δηλαδή της επανεξέτασης της δομής των προϊόντων υπάρχει, το έχουμε τονίσει από την, αρχή, από την αρχή και ήδη είμαστε μάρτυρες αλλαγών και αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν. Καταρχάς. Κατά δεύτερο, για τα ωφελήματα, τις ενισχύσεις, τα επιδόματα κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο ε, ασφαλιστικό, είναι και συνταξιδετικό το θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το πίσω μέρος των βιβλίων, γιατί οι περισσότερες νέες διευθετήσεις εξαρτώνται από τη συνεισφορά στο ταμείο, είτε το θέλουμε είτε το όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για τα παλιά λοιπόν, σε δύο επίπεδα δουλεύουμε. Πρώτον, αναλύουμε την φρεγγιότητα των συνταξιδοτικών ταμείων και ελπίζουμε ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς θα δώσουμε στα ευρωπαϊκά πολιτικά θεσμικά όργανα γνωμοδότηση για το πώς θα δημιουργηθεί πλαίσιο για την ανάλυση της βιωσιμότητας των μακροπρόθεσμων υποσχέσεων. Και αυτό πρέπει να είναι διαφανές, με διαφάνεια να γίνει, για να το αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά. Και κάνουμε stress test, τεστ αντοχής στα συνταξιδοτικά ταμεία, ε, στα τέλη αυτής της χρονιάς και οι υποσχέσεις που θα δίδονται μετά θα είναι μέρος του αποτελέσματος των stress test. Ευχαριστώ. Παύλο Σάινς. Παύλο Σάλμπα μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους τρεις προέδρους για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση γενική. Όποιος θέλει την απαντάει. Ε, Υπάρχει μεικτή επιτροπή των τριών εποπτικών ε, αρχών και εξέδωσε ε, μία έκθεση με συστάσεις που ε, ήταν συμφωνή με τις προτάσεις του Επιτρόπου Χίλ με σκοπό τη δημιουργία περισσότερης απασχόλησης. Ποια είναι τα πεδία δράσης που βλέπετε, ποια περισσότερα πεδία δράσης, πού θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση περισσότερη για να δημιουργηθεί περισσότερη απασχόληση. Και επιστρέφω, επανέρχομαι στις τιτλοποιήσεις στην Ευρώπη και για το πώς χρησιμοποιούνται. να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει τη συγκεκριμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ύπαρξη μιας ενιαίας κεφαλαιακής αγοράς, ενιαία κεφαλαία αγορά. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε ποιους πυλώνες πρέπει να εδράζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ε, κεφαλαίων τιτλοποίησης και και ποια είναι τα βήματα για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ευχαριστώ. Ο Στίβεν, εν συντομία να απαντήσω και για το θέμα της τιτλοποίησης και για το ευρύτερο που, ε, θέμα που θίξατε για την Ένωση Κεφαλαγορών της Ευρώπης. Πράγματι, οι τρεις εποπτικές αρχές ως προς την τιτλοποίηση δούλεψαν από κοινού και ε, μείναμε προσιλωμένοι στη συνέπεια του πλαισίου τιτλοποίησης στα διάφορα είδη νομοθεσιών. Τα περασμένα χρόνια έχετε δει ότι έχουν υπάρξει νέα προαπαιτούμενα τιτλοποιήσεων ως στην νομοθεσία για την ασφάλιση των τραπεζών και τις κεφαλαιακές προϋποθέσεις, τη κεφαλαιακή επάρκεια, όλοι θα ωφεληθούν από περισσότερη συνέπεια, περισσότερο streamlining, ευθυγράμμιση της νομοθεσίας, η οποία να ε, γυρνάει γύρω από τους ίδιους ανοιολογικούς άξονες. Και υποβάλαμε αυτή την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιευτεί και στη δική μας ιστοσελίδα. Είναι δημόσια γνώση. Ο Ανδρέα θα μιλήσει περισσότερο για το θέμα της τίτλοποίησης και ε, κυρίως της κεφαλαιακής επαρκίας, όμως από πλευράς ΕΣΜΑ Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά πάνω στο πεδίο των αποκαλύψεων και τη διαφάνεια. Ένα από τα προβλήματα τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση ήταν ότι οι επενδυτέ δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν την ποιότητα των διαφόρων χαρτοφυλακίων γιατί δεν υπήρχε αρκετή διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της αγορά τυπλοποίηση και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αλλά δεν ήταν και το πιο εύκολο εγχείρημα γιατί προκύπτουν διάφορα προβλήματα. Έχουμε αρκετούς πόρους για να φτιάξουμε μια επαρκή ιστοσελίδα που ε, θα παρέχει την τηλεοποίηση τη διαφάνεια για τις τηλεοποιήσεις. και από εκεί και πέρα πώς θα στηρίξουμε την Ένωση Ευρωπαϊκών Κέφαλαι Αγορών, πώς θα στηρίξουμε την ανάπτυξη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια σήμερα να απαντήσουμε, αλλά πρέπει να προχωρούμε βήμα προς βήμα, να εξετάζουμε τα επιμέρους στοιχεία των ευρωπαϊκών χρήματα αγορών και χρηματοπιστωτικών αγορών να ανοίξουμε και να αναπτύξουμε ορισμένους διάβλους πέρα από το διάβλο της τιτλοποίησης, να ανοίξουμε το διάβλο του, crowdfunding αλλά και το διάβλο του asset management, της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού μεταξύ άλλων. Δηλαδή αυτά τα μονοπάτια θα τα κάνουμε λεωφόρους και ε, να έχουμε συνεπή υλοποίηση των υφιστάμενων κανονιστικών μεταρρυθμίσεων. Ξέρετε πολλές από τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις είχαν ε, ε, επινοηθεί στο πλαίσιο πλαίσιο της σταθερότητας και της προστασίας. Ωστόσο, πολλά έγιναν τα, τα περασμένα χρόνια και πέρσι για το Single Rule Book, για τους ενιαίους κανόνες και πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά, να τα πάμε ένα βήμα πιο πέρα για να υπάρχει συνέπεια στα 28 ε, κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Πίτερ Ζήμων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε η κυρία Φερέρα. Ήδη πριν από δύο εβδομάδε αποφασίσαμε τα του προπολογισμού του 2016 και μας εξηγήσατε τι συνέπειες έχει η χρηματοδότηση που έχετε αυτή τη στιγμή και ε, βεβαίως εμείς ως Κοινοβούλιο είχαμε ζητήσει την αύξηση της χρηματοδότησής σας αλλά εσείς μας είπατε πως ακόμα και αυτό δεν είναι το 100% των όσων θα θέλατε. Αναφερθήκατε παραδείγματο χάρη συλλογή δεδομένων και τα συστήματα πληροφορική. Μα πώς θα κάνετε τη δουλειά σας όταν υπάρχουν ελλείψεις ήδη στη συλλογή των ε, δεδομένων. Και υπάρχει ένα ερώτημα που θα ήθελα να απευθύνω και στους ε, τρεις σας. Εάν ναι, παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο χρηματοδότησής σας, μπορείτε να μας πείτε πώς εκτιμάτε μακροπρόθεσμα το εάν θα μπορείτε να επιτύχετε τα όσα σας έχουμε αναθέσει ως αποστολές όπως αναμένει ο φορολογούμενος και το Κοινοβούλιο ή να μας πείτε ποια χρηματοδότηση απαιτείται για κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο μου ερώτημα επίσης πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και το ερώτημα είναι ποιος τα πληρώνει αυτά. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη και των τριών σας. Τι άποψη έχετε για την πρόταση της ΕΚΟΝ που λέει να μην ε, έχουμε συνεισφορές ε, των εθνικών αρχών και των κρατών μελών, αλλά να χρηματοδοτηθείτε από τέλη που θα επιβάλλονται στους συμμετέχοντες στην αγορά ή εναλλακτικά να έχουμε μια μεικτή χρηματοδότηση. Τέλη των ε, συμμετεχόντων και συνεισφορές αυτόν τον προπολογισμό της Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν. Κάποιες ε, αντιδράσεις. Πρώτον και όπως ίσως ε, γνωρίζετε το σύστημα χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση από τον Επίτροπο Χίλ, ε, είναι τμήμα της εντολής του και βεβαίως εξετάζει ακριβώς την βελτίωση της χρηματοδότησης των τριών αρχών. Πράγματι όπως επισημάνατε είναι σημαντικό να μειωθεί και να καταργηθούν οι συνεισφορές των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των εθνικών αρμοδίων αρχών και ο λόγος είναι πως είναι πάρα πολύ άδικο και δεν είναι και λογικό γιατί περισσότερα κονδύλια για τις αρχές σημαίνει ε, λιγότερα κονδύλια για τις εθνικές αρχές και αν δείτε την νομοθεσία που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο πολύ μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυξάνονται οι αρμοδιότητες, οι υποπτικές και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπα λοιπόν, τώρα επαφίεται στον Επίτροπο να τα προχωρήσει αυτά να δυνατόν πιο γρήγορα. Σύντομα λοιπόν. Δεν πρέπει να υποτιμάμε ότι σε τελική ανάλυση η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά η εφαρμογή του επίπεδου 2 και το να γίνει με τρόπο σωστό είναι η μισή δουλειά και βέβαια στο να μην έχουμε επαρκής ε, πόρους υπονομεύει συνολικά τους στόχους ε, της ε, ρυθμιστικής αυτής μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Όχι. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Ποιος? Η Κέι Σουίνμπρον. Ευχαριστώ. Έχω και δεύτερη ερώτηση. Θα κάνω την ερώτηση που ε, δεν θεωρούσα ότι είχα χρόνο να κάνω. Απευθύνομαι στον κύριο Ενρία για το θέμα του συστήματος ε, του ε, CSDR με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε γιατί ξέρετε πως εμείς πάντα ήμασταν υπέρ της επαρκούς κεφαλαιακής κάλυψης για τις πιο επικίνδυνες δραστηριότητες και άρα δεν δεχόμασταν τον πλήρη διαχωρισμό των συστή από, ε, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θεωρούμε πως θα πρέπει να προσθεθούν όσον αφορά την ρευστότητα για να αξιολογηθεί πλήρως ο κίνδυνος. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς ε, προχωρούν τα πράγματα σε αυτό τον φάκελο και πώς ακριβώς ε, ισορροπείτε τις πολύ υψηλέ απαιτήσει των εποπτικών αρχών των κρατών μελών που εποπτεύουν τους μεγάλους αυτούς οργανισμούς για το κείμενο αυτό επίπεδου 2. Και επίσης για ένα χρονοδιάγραμμα θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, ερώτηση. Ήταν δύσκολο το θέμα, όπως ξέρετε. Έγινε μια διαβούλευση και προτείναμε κάποια κριτήρια ακριβώς για να δούμε ποιες θα ήταν οι επιπλέον κεφαλιακές απαιτήσεις ε, για τα κεντρικά αποθετήρια που παρέχουν τέτοιες ε, τραπεζικές υπηρεσίες και λάβουν πάρα πολλές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ε, διαβούλευσης και τώρα βεβαίως ε, οριστικοποιούμε την τελική μας πρόταση και ελπίζω πράγματι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ήδη εντός του μηνός ή το αργότερο το επόμενο μήνα. και ευχαρίστω βεβαίω και διμερός ε, να το δούμε αλλά το βασικό είναι να έχουμε όπως είπατε αυτές τις επιπρόσθετες ε, απαιτήσει ρευστότητα. Ένα βασικό σημείο βεβαίως αφορά και τα νομίσματα και το τι γίνεται με το νόμισμα με το οποίο λειτουργεί το κάθε κεντρικό αποθετήριο αξιών και το σε ποια νομίσματα έχουν εκτεθεί. Εκεί πέρα εστιαζόμαστε τώρα. Σας ευχαριστώ. Η Εύα Παούνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες οι συμμετέχοντες της αγοράς και οι πολιτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες τους για την πρόταση της ε, ΕΣΜΑ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΜΥΦΙΤ 2 ότι δηλαδή οι συνεργασόμενοι θα πρέπει να δημοσιοποιούν τις ε, τιμές ε, για το χρέος και μάλιστα το κατόφλι για το οποίο, από το οποίο ένα ομόλογο θα υπόκειται σε αυτές τις απαιτήσει ε, δημοσιότητας ε, είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν ενισχύει την ε, ρευστότητα και βεβαίως ο κίνδυνος θα είναι πώς θα μπορούσαν να στεγνώσουν οι αγορές του χρέους ειδικά σε μια εποχή στην οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή η ρευστότητα οπότε βεβαίως το ερώτημα είναι και ποια μόλγα είναι ε, ρευστά και πια όχι αυτή την στιγμή. Θεωρείτε λοιπόν πως θα μπορέσετε να, καταλήξετε, να καταλήξετε σε ένα ε, σύστημα το οποίο θα έχει βρει την ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και ρευστότητα και στην περίπτωση στην οποία δεν γίνει αποδεκτό αυτό ποιες επιλογές θα προτείνετε στον κλάδο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Όπως ε, σωστά επισημάνατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του MIFID 2 και του MIFID η διαφάνεια στην αγορά ομολόγων και η ΕΣΜΑ πάντα ε, θεωρούσε πως η διαφάνεια και η ρευστότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική σε σχέση με τις μετοχές. Οπότε όταν υπάρχει διαφάνεια στην αγορά ομολόγων πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός και να γίνει στοχευμένα γιατί αν δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την ε, ρευστότητα. Ειδικά στα σημεία εκείνα στα οποία είναι ήδη περιορισμένοι. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχει τύχει ιδιαίτερη προσοχή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό. Εγώ θα έλεγα το εξή. Η πρόθεση του νομοθέτη στην ΜΥΦΗ 2 και την ΜΥΦΙΡ είναι να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στην αγορά ομολόγων, καθώ η υπόθεση είναι ότι αν αυτό γίνει προσεκτικά μπορεί να οδηγήσει η διαφάνεια και σε περισσότερη ρευστότητα, γιατί οι επενδυτέ θα εμπιστεύονται περισσότερο την αγορά και θα μπουν σε αυτήν ε, το εξάζουμε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικά. Υπάρχει ακριβώς και η γνωστή συζήτηση για την κόφια και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τελικά πως μόνο ένα μικρό κομμάτι της αγοράς ομολόγων θα θεωρηθεί ότι έχει ρευστότητα και άρα θα υπόκειται σε αυτές τις απαιτήσεις διαφάνειας. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα γύρω στο 1-5% της αγοράς ομολόγων θα καλύπτεται από αυτές τις απαιτήσεις διαφάνειας. Εάν παρελπίδαν. Όταν δημιουργηθεί το σύστημα υπάρχουν αρνητικές ε, επιπτώσεις ή κάποιες ε, συνέπειες ε, οι οποίες μίες και μένες, τότε θα επανεξάσουμε το σύστημα και θα υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα της έκον για παρόμβαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα της κυρίας Χούμπνερ. Με, με κοιτάτε. Κύριε Βαϊτσέκερ, ε, για το θέμα της αναζήτησης αποδόσεων που θεωρώ πως είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους των χαμηλών επιτοκίων. Το πρώτο μου ερώτημα είναι ποιες ενδείξεις έχετε για το εάν οι αναζητήσεις ε, αποδόσεων ε, αυτή τη στιγμή είναι το βασικό κίνητρο ασφαλιστικών εταιριών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Και δεύτερον, κατά πόσον ε, θεωρείτε πως αυτό έχει ως κίνητρο την έκπτωση που υπάρχει στην πλευρά της ευθύνη. Θεωρείτε παραδείγματο χάρη πως ε, το μεγάλο αυτό ποσοστό έκπτωση μας δίνει μια στρεβλωμένη αξία του επίπεδου φερεγγιότητας των ασφαλιστικών εταιριών και τι θα πρέπει να κάνουν σε αυτή την περίπτωση οι εποπτικές αρχές. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά επίσης τις εκθέσεις που έχει συντάξει για κινδύνους και αδυναμίες. Λέει πως οι εποπτικές αρχές πρέπει να, δουν μια, να έχουν μια ολιστική άποψη και να ερμηνεύουν ευέλικτα βεβαίως ε, τα των ασφαλιστικών ταμείων. Πολύ ωραία έκφραση, αλλά τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά ακριβώς αυτές τις εκτό που αναφέρθηκαν. Θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για, το, ε, για να επιτύχουν το επίπεδο φερεγγιότητας, ε, ένα διαφορετικό τρόπος υπολογισμού του. Με άλλα λόγια, τι ακριβώς εννοείται εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για το κυνήγι των ε, αποδόσεων, ε, το κοιτάμε και από ποιοτική και ποσοτική πλευρά. Την πλευρά την ποιοτική, τα νούμερα που έχουμε τώρα, προσπαθούμε να βρούμε κάποια νούμερα τα οποία θα είναι θα εκφράζουν την πραγματικότητα και δεν δείχνουν πως υπάρχει μια τεράστια απόκληση σε σχέση με το παρελθόν. όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείε όμως στην ποσοτική αποτίμηση που κάνουμε βλέπουμε οπωσδήποτε μια αύξηση κάποιων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν ήταν παραδοσιακές θα έλεγα για τον κλάδο των ασφαλιών βλέπουμε έκθεση σε πιστώσεις είτε μέσω τραπεζών είτε απευθείας επίσης οι υποδομές αυξάνονται και το βλέπουμε αυτό. Ότι δηλαδή θα έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα νούμερα για να είμαστε σαφείς. Όσον αφορά το θέμα, όπως είπαμε, των αδυναμιών και τι συμβαίνει στο πλαίσιο της οδηγίας για τη φεργιότητα 2, οπωσδήποτε είναι μέρος του υφιστάμενου καθεστώτος. Ήταν κάτι το οποίο το φέραμε στη φεργιότητα 2 από το Omnibus 2 για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα κύκλικα στοιχεία με έναν τρόπο που θα είναι πολύ πιο συνεπής με την αγορά. Οπότε το αναμενόμενο, το μελλοντικό επιτόκιο είναι ε, κάτι το οποίο υπάρχει και είναι σαφές ε, στον Omnibus 2 πως ε, το μελλοντικό αυτό επιτόκιο δεν μπορεί να αλλάζει συνεχώς. Οπότε πρέπει να είναι κάτι το σταθερό για να μην έχουμε ακριβώς αυτή την κυκλική συμπεριφορά και την υπερβολική αναταραχή. Τώρα έχουμε έρθει σε επαφή με τις ε, εταιρείες αυτές και είναι μέρος ε, της προετοιμασίας μας και η απόφασή μας είναι πως όταν θα τεθεί ενισχύ το καθεστώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία είχαν γίνει για τον αρχικό καθορισμό του στήματος αυτά τα οποία χρησιμοποιήσετε και εσείς για να λάβετε την αρχική σας απόφαση ε, για το Omnibus 2, αλλά ταυτόχρονα εξετάζουμε και την μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται όπως είπαμε και για το DIRFAR και σκοπεύουμε να έχουμε και άλλη μια ευρύτερη διαβούλευση το 2016 για να αναθεωρήσουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε ήδη εδώ και χρόνια πρέπει να λάβουμε υπόψη τι παράγοντες χρησιμοποιούμε, τι συντελεστές πώς πρέπει να αξιολογήσουμε τις πραγματικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις και τον πληθωρισμό και οπωσδήποτε να αποφύγουμε το να υπάρχουν ε, κάποιες ε, συνέπειες ε, οι οποίες δεν ήταν αυτές οι οποίες θα θέλαμε. Τώρα όσον αφορά το στοιχείο αυτό της ολιστικής αντιμετώπισης των αδυναμιών και της φερικιότητας. Κοιτάξτε, από την πλευρά των ασφαλιών έχουμε ήδη κάποια στοιχεία που υπάρχουν στο αριθμιστικό καθεστώς ε, όσον αφορά τα μεταβατικά στοιχεία, τις ε, μεταβατικές ε, περιόδους, πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίζει αυτό η τα κτλ. Στην πλευρά των στεξιωτικών ταμείων τώρα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο ανάλυσης της φερεγγιότητας. Εξετάζουμε, όπως είπαμε, την ολιστική αυτή αντιμετώπιση Τη φερικαιότητας των εξοδοτικών ταμείων για να είμαστε πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι σαφής. Αν δει κανεί τι μακροπρόθεσμε υποχρεώσει ε, πιο ρεαλιστικά, δύο πράγματα μπορεί να γίνουν να, για να χρηματοδοτηθούν. Είτε αυξάνονται οι εισφορές, είτε μειώνονται οι παροχέ. Ε, δεν μπορεί να γίνουν θαύματα και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως εμείς λέμε ε, ότι πρέπει να μην είμαστε ευέλικτοι. Όχι, είναι πολύ μακροπρόθεσμες αυτές τις μέρες, αλλά για να μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις πρέπει να έχουμε αριθμούς και μια ρεαλιστική αξιολόγηση και αυτό ακριβώς θεωρούμε εμείς μια ρεαλιστική άποψη όσον αφορά τη φερεγγιότητα των στεξιωτικών ταμείων. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Πέτερ, ευχαριστώ. Η τελευταία μου ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Ενερία. Στις 14 Απριλίου φέτος είχαμε εδώ πέρα τον κύριο Φακάση, τον εκτελεστικό διευθυντή και συζητήσαμε τα σχέδια εκτελεστικών προδιαγραφών ε, σύμφωνα με το άρθρο 36 και βεβαίως ε, το ερώτημα ήταν η μικρή οικία αξιολόγηση σε σχέση με τους μεγάλους γιατί βλέπουν εκεί πέρα το ποιο επίπεδο φερεγγιότητας ε, ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση του κάθε οικοξιολόγηση. Βεβαίως το θέμα εδώ πέρα είναι πως ε, το εάν μεταφράζονται αυτές οι αξιολογήσεις άμεσα σε κάτι ή εάν εξαρτώνται από τον κάθε οίκο αξιολόγησης ε, για το εάν θα μπορεί παραδείγματος χάρη να δώσει προσεχώς ένα 3α. Δηλαδή, εάν ε, ισχύσει λοιπόν αυτό το οποίο είπατε, δεν θα, δεν θα μπορούσαν να μπουν νέες μικρές εταιρείε στον κλάδο γιατί θα έπρεπε να έχουν του έναν ελάχιστο αριθμό αξιολογήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι έχετε κάνει για να βελτιωθεί εδώ πέρα η κατάσταση γιατί κατά την ε, άποψή μας υπάρχει ένα σαφές ε, μειονέκτημα για τις, μικρές αυτές, για τις μικρούς οίκους αξιολογήσεων και ακριβώς η κρίση κατέδειξε πως η κυριαρχία των υφιστάμενων μεγάλων ε, δεν είναι υγιής. Ένα άλλο ερώτημα για τις τεχνικές προδιαγραφές και το πώς θα ληφθεί υπόψη η αρχή ότι θα πρέπει να έχουμε μια περίοδο χάριτος τις ε, μικρότερες ε, τις μικρότερες οίκους αξιολόγησης. Τι έχει γίνει με αυτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Ανδρέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ήταν ένα πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί την Κομισιόν. Από άποψη προληπτική, στόχος και ανησυχία μας είναι να γίνει μια στεναρή αξιολόγηση των κινδύνων. Και βεβαίως, όσο πιο στεναρός είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση, τόσο πιο σίγουρος είναι. Και αυτό σημαίνει βέβαια δυσκολία για τις νεοδημητές ε, αυτές, ε, τους οργανισμού αυτούς τους οργανισμούς αξιολόγησης, κυρίως ε, ε, για την πρώτη τάξη αξιολόγηση. Δεν είναι βέβαια αδύνατον να αναπτύξουν αυτή την εργασία, αλλά είναι αυτή τη στιγμή υπό κάποιους περιορισμούς. Επίσης, προσπαθούν να βρουν τη σωστή ισορροπία και άραγε ισχύει αυτή τη στιγμή μία περίοδος χάριτος κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτό το στοιχείο που προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία και αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η συνεπία ανάμεσα σε αυτήν την στάνταρ μεταχείριση των ε, CRAs για τους στόχους της που υπήρξε ευθυγράμμιση ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις και θέλουμε να βρούμε και να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι μια περίοδος χάρτος ήταν η σωστή προσέγγιση. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Το ίδιο, η ίδια περίοδος χάρτος θα ισχύσει και για το Solvency 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Ανδρέα, Γκάμπριελ και Στέβεν για αυτή την πολύ πολύ πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Εγώ δεν μπορώ να συνοψίσω τα πολύ σημαντικά θέματα που προέκυψαν και επί των οποίων θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, να συζητούμε. Μόνο να υπογραμμίσω ε, μία τελική παρατήρηση που αφορά τους πόρους ε, και νομίζω ότι όλα όσα μας είπατε και βέβαια και η λογική και το πνεύμα των ερωτήσεων δείχνει ότι οφείλουμε να σας στηρίξουμε για αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο και να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα το οποίο να είναι κατάλληλα χρηματοδοτούμενο. Θα συνεχίσουμε φυσικά το διάλογό μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. So I will go quickly to the announcement and then to Γρήγορα τις ανακοινώσεις και μετά στο υπερνάμε στις ψηφοφορίες. Να σας θυμίσω την συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής την επόμενη πέμπτη το πρωί από τις 10 μέχρι τις 12.30 κατά τη διάρκεια της οποίας μαζί με την Επιτροπή ΤΑΚ θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψε με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον Πιέρ Μοσκοβισή και την Μάργαρετ Βεστάγκερ για την θέματα φορολογίας προφανώς. Και επίση να σας πω ότι αύριο από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού, της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οπότε στη διάρκεια του μεσημεριού, του μεσημεριανού διαλύματος θα τακτοποιηθεί η αίθουσα έτσι ώστε να υποδεχτούμε του προσκεκλημένους μα και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσια διάταξη, έγκριση του σχεδίου προγράμματο των συνεδριάσεων τη Επιτροπή μα για το 2016. Έχετε πάρει το κείμενο, θα έλεγα ότι αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι εγκρίνεται αυτό το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο είναι το σημείο 8, νέα διαβούλευση. Πολύ καλά, ναι, για το σημείο 8 διακόπτει ο Πρόεδρος. Όπως γνωρίζετε, έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία επί της οδηγίας κατανομής ε, ε, ασφαλίσεων ε, είναι, το άλλαξε και ο τίτλος τώρα δεν έγινε πια διαμεσολάβηση θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λάγκη και τη διαπραγματευτική μας ομάδα και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε σύμφωνα με το κανονισμό μας αλλά θα ήθελα εξ ονόματος του κύριου Λάγκη να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλτς ναι, Ευχαριστώ κύριο Λάγκεν είναι καθοδόν προς Βρυξέλλες αλλά έχει κολλήσει στο ποτηλιάρισμα και μου ζήτησε να πω λίγα λόγια. Θα είμαι σύντομος. Ε, η πρώτη συμβασμού για μια νέα ρύθμιση των ασφαλιστικών υπηρεσιών οπωσδήποτε είναι κάτι που μπορεί να στηρίξει. Αυτό το οποίο ζητάμε εμείς ως Κοινοβούλιο δηλαδή να υπάρχουν ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και για την ενημέρωση και για απαιτήσει ε, ε, προσόντων και καταγραφής ε, των εταιριών εκπληρώνονται. Νομίζω πως αυτό είναι ιδιαίτερος θετικό. Μπορούμε να πούμε και άλλα πολλά και διάφορα βεβαίως. Αλλά νομίζω πως θέλουμε να ψηφίσουμε. Ο Βέρνερ Λάγκεν επίσης μου είπε, μου ζήτησε ρητός να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και τους ε, συνεργάτες της γραμματείας της ε, ΕΚΟΝ, τον Γιονιφανές και την Σατάσα Μαλίκα και ζητάει να ε, συμφωνήσετε με αυτή τη συμβιβαστική πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη γραμματεία μαζί με τον κύριο Λάγκη για την εξαίρετη στήριξη, υποστήριξη που μας προσέφερε η επιστολή του Συμβουλίου έχει κυκλοφορήσει και οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτα θα κάνουμε μια δοκιμή. Δοκιμαστική ψηφοφορία άρχεται. Τέλος. Εντάξει, λειτουργούν όλα τα μηχανήματα, οπότε μπορούμε τώρα να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Vote is closed. Πέρας. 31 ε, υπέρ, 4 αποχές. Πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως και τώρα θα πρέπει να επικυρώσει να κυρώσει μάλλον αυτή την ε, συμφωνία της πρώτης ανάγνωση όσον αφορά την οδηγία περί ε, κατανομής ασφαλίσεων. And I no. Okay, I will start, uh, uh which is scrutiny of delegated. Και τώρα θα εξετάσουμε την κατεξιδότηση πράξη και τα εφαρμοστικά μέτρα για τα PRIPS. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, για τα μέτρα που προετοίμασαν οι ΕΣΑΣ και η Κομισιόν και όπως ξέρετε αποδίδουμε μεγάλη σημασία στα μέτρα αυτά. Σήμερα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα πρίψη ενημερωτικά έγγραφα για επενδυτικά προϊόντα, βασικά ενημερωτικά έγγραφα για επενδυτικά προϊόντα, μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και βεβαίως απαιτείται διατομεακή συνεργασία και αυτό είναι και το τέλειο παράδειγμα, γι' αυτό ήταν σωστό να δημιουργηθεί μεικτή επιτροπή των τριών ΕΖΑ. Ο κανονισμός των PRIPS επίσης ε, δίνει δυνατότητα παρέμβασης στα προϊόντα, ε, στα ασφαλιστικά. Ε, γι' αυτό σήμερα θα θέλαμε όλος ιδιαίτερα να συζητήσουμε το, έγγραφο, το τεχνικό έγγραφο που προετοιμάστηκε από τη Μικτή Επιτροπή των Τριών ΕΖΑ στις 30 Ιουνίου όσον αφορά το κόστος της αποκάλυψης καθώς και τα βασικά ενημερωτικά έγγραφα για τα επενδυτικά προϊόντα. Ένα τεχνικό έγγραφο συζήτηση που στόχο έχει να προσφέρει στου ενδιαφερόμενου την ευκαιρία να σχολιάσουν ορισμένε συγκεκριμένε τεχνικέ πτυχέ που σχετίζονται με την απόδοση κινδύνου και την πληροφορία περί κόστου. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στι 17 Αυγούστου και αυτή τη στιγμή οι ΕΖΑΣ αξιολογούν τις πληροφορίες που συνέλεξαν και μετά θα ασχοληθούμε με το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών λεπτομεριών ε, προδιαγραφών που θα ε, υποβληθεί μέχρι 31 Τρίτου του 2016 στην Επιτροπή μας. Έχουμε λοιπόν εδώ λεπτομέρειες να εξετάσουμε και να ακούσουμε και την άποψη των ενδιαφερόμενων φορέων όπως προς αυτό και πάλι θα καλωσορίσω τον Στέβεν Μέιτζορ που θα πάρει το λόγο εξ ονόματος της Μικτής Επιτροπής, τον ΕΖΑ, καθώς και τον κύριο Κέτνερ που είναι ο υπηρεσιακός επικεφαλής της ε, μονάδας ΒΙΣΜΑ. Σύντομη εισήγηση θα ακούσουμε τώρα. Παρακαλώ να μην πάρετε πάνω από 10, maximum 15 λεπτά και για τα δύο και μετά η διαπραγματευτική ομάδα για τα πρίψε θα υποβάλει ερωτήσεις προς εσάς. Κυρία Στίβεν. Α, όχι. Η Επιτροπή πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις εργασίες μετά την υιοθέτηση του κανονισμού για πακεταρισμένα επενδυτικά προϊόντα με βάση τη λιανική και τις ασφάλειες, PRIPS. Η ιδέα είναι βασική και απλή. Οι αποταμιευτές στην Ευρώπη χρειάζονται σαφή πληροφόρηση για το κόστος που πληρώνουν και το κίνδυνο που αναλαμβάνουν όταν επενδύουν. Το KID, το βασικό έγγραφο πληροφόρησης, θα αποτελέσει για πρώτη φορά κοινό πρότυπο ενημέρωσης για όλα τα είδη επενδυτικών προϊόντων που βασίζουν την απόδοσή τους ε, όχι σε, στις επιδόσεις που ε, κερδίζει άμεσα ο επενδυτής. Έχουμε συνδυασμό χρηματοπιστωτικών εργαλείων, έχουμε τιμές αποδόσεων και τιμές αναφοράς για να δούμε ε, πόσο ε, παίρνουν ακριβώς οι ε, επενδυτές, οι retail επενδυτές. Και όλοι μετά το 2016 θα πρέπει να συμμορφούνται με αυτούς τους κανόνες. Το PRIPS θέλει να μην υπάρχει περιπλοκότητα, να μην υπάρχει δύσκολη ιδιόλεκτος και το ΚΙΔΙΟ, το βασικό πληροφοριακό έγγραφο για αυτά τα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται στους αποταμιευτές, τους πολίτες να μην ξεπερνά τα, τις τρεις σελίδες. Έχουμε πολύ πιο λεπτομερείς κανόνες για το KID, το Key Information Document και ο Στίβεν θα σας ενημερώσει για αυτές τις εξελίξεις. Ε, θα ήθελα να σταθώ δύο λεπτά για να εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι έχουμε κάνει για να στηρίξουμε τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και ε, για να δούμε ότι εφαρμόζονται οι κανόνες για το KID. Για να είναι χρήσιμο το KID το βασικό πληροφοριακό έγγραφο στους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει μια σύμβαση για τη διενέργεια μιας μελέτης δοκιμής καταναλωτικής. Δηλαδή ήταν σχεδιασμένη η μελέτη έτσι ώστε να μάθουμε ποιο τρόπο παρουσίασης της πληροφόρηση καταλαβαίνουν καλύτερα οι καταναλωτές και πώς, τι τους βοηθάει να συγκρίνουν τα διάφορα ε, επενδυτικά ε, καταναλωτικά προϊόντα. Έγινε αυτή η μελέτη σε 10 κράτη-μέλη και ε, είχαμε προσεκτική επιλογή για ευρεία γεωγραφική κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης τέτοιου είδους αγοράς επενδυτικών προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, για να είμαστε βέβαιοι ότι η διαμόρφωση και η μορφή ε, του βασικού πληροφοριακού εγγράφου δουλεύει πατού, έχουμε τρία είδη προϊόντων, δομικά προϊόντα, ε, συμβάσει, συμβόλαια ασφάλισης ζωής με διάφορες επενδυτικές επιλογές μεταξύ άλλων. Έχουμε ε, τρεις βασικές επικεφαλίδες, αν θέλετε, τρεις κατηγορίες ε, επενδυτικών προϊόντων. Και ε, ως προς την παρουσίαση κεντίνου και σενάριο επιδόσεων και ενημέρωση για το κόστος, για αυτά τα θέματα οι καταναλωτές προτιμούν ε, απλούς δείκτες συνοπτικούς και περιληπτικούς. Δεν θέλουν υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες και υποκατηγορίες. Και ε, η παρουσίαση του κινδύνου είναι μεγάλη πρόκληση για το ΚΙΝΤ. Ένας δείκτης βασικός ε, αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα οι καταναλωτές. Αυτό είδαμε. Δηλαδή ένα προϊόν ταξινομείται σε μια κατηγορία κινδύνου από το 1 μέχρι το 7 σε, ε, ε, και αυτό εξαρτάται με το συνολικό κίνδυνο. Δεν έχουμε επιμέρους ανάλυση κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο πίστοσης, εμπιστοσύνης. Δεν έχουμε τέτοιου είδου επεξηγήσεις διότι οι καταναλωτές δεν τις προτιμούν και προτιμούν τα σενάρια σε σχέση με το μέλλον. Οι μελέτες έδειξαν ότι τα σενάρια επιδόσεων, ότι το σενάριο α θα έχει τυχή απόδοση, το β, το γ κτλ. Ε, είναι αυτά που προτιμούν οι καταναλωτές έχοντας αφαιρέσει στο τέλος βέβαια ε, τα κόστη. Και δεν θέλουν οι καταναλωτές ε, γραφήματα, αλλά προτιμούν γραφικές παραστάσεις. προτιμούν πίνακες και όχι γραφήματα δυσκολεύονται να κατανοήσουν διαφορετικά είδη τους, δηλαδή τα έκτακτα, τα μόνιμα, τα τρέχοντα και το πώς διαχωρίζονται όλα αυτά μεταξύ τους. Οι θα θέλουν μια απλή παρουσίαση και βασίζονται γενικά στη, στο συνολικό νούμερο του πόσο θα είναι το κόστος για το χ προϊόν και όχι πώς επιμερίζεται αυτό το κόστος το κόστος. Η μελέτη θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο και με χαρά θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και άλλες ερωτήσεις για τη μελέτη ήδη από σήμερα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος. Και εμείς ευχαριστούμε να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μάιζορ. Στίβεν, παρακαλούμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι. Θα κάνω μια σύνοψη της δουλειάς που έχουμε κάνει για τα περίψε εμείς οι ε, τρεις εποπτικές αρχές και υπεύθυνο από την ΕΙΟΠΑ θα είναι εδώ για να απαντήσει στα ερωτήματα που κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψουν ε, την ε, επόμενη ώρα. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, με χαρά δράτω με τις ευκαιρίες ως ε, συμπρόεδρος τη Επιτροπής των Τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για να ενημερώσω τις Επιτροπής σα για τη δουλειά που κάναμε για τα τεχνικά κανονιστικά πρότυπα για το ΠΡΙΠΣ, το βασικό έγγραφο ε, το βασικό πληροφοριακό έγγραφο, το KID, είναι η πιο σημαντική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, γιατί ενδιαφέρει και τους επενδυτές και ενισχύει την προστασία του καταναλωτή. Ε, νομίζουμε ότι αυτό θα είναι το πιο ορατό στοιχείο ε, που θα κάνει τον Ευρωπαίο πολίτη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει πραγματικά τη δουλειά που κάνουν οι τρεις εποπτικές αρχές. Ξεκινήσαμε το 2012 και εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας μετά την πολιτική συμφωνία τον Απρίλιο του 2014 για τον κανονισμό για τα PRIPS και θέλω να τονίσω την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί ε, η οποία είναι υπέρ της διαφάνειας. Έχουν δημοσιευτεί ε, δύο ε, εκθέσεις και έχουν διοργανωθεί πάρα πολλά πάνελ με συμμετοχή ειδικών πανεπιστημιακών και εκπροσώπων του κλάδου. Στη συνέχεια θα έχουμε διαβούλευση για τις κανονιστικές τεχνικές προδιαγραφές το Νοέμβριο και Έχουμε εκτεταμένη άσκηση προτιμήσεων των καταναλωτών, την οποία διενήρξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την οποία σας μίλησε μόλις τώρα. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι επιλογές ε, πολιτικής ε, ε, ενσωματώνουν το feedback από τους καταναλωτές. Το ποσοστό επιτυχίας θα εξαρτηθεί από την παρουσίαση αλλά και από το περιεχόμενο του εγγράφου, του βασικού πληροφοριακού εγγράφου θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στα RTS, τα technical standards, τα κανονιστικά που συνάδουν με αυτές τα προαπαιτούμενα και όλα αυτά να γίνουν μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2016. Είναι μεγάλη η δρασή του RTS αυτού και των τεχνικών προδιαγραφών για την αναθεώρηση και επανεξέταση του κίνητου, του βασικού πληροφοριακού εγγράφου. Θεωρούμε ότι αξίζει να, να ε, έχουμε τις ίδιες προθεσμίες και το συνολικό πακέτο να το παραδοθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Επισήμω λοιπόν θα έρθουμε σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους συνομοθέτες, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, εν συντομία ε, ζητώντας ίδιες προθεσμίες και για τα δύο. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για τις τρεις εποπτικές αρχές και να υπογραμμίσω ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι τελικές αποφάσεις για το τι θα βάλουμε στο επικείμενο έγγραφο διαβούλευσης. Ωστόσο, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να δώσω κάποιες ενδείξεις για το ε, προς τα που θα κατευθυνθούμε και ευχαριστώ θα λάβουμε υπόψη μας δικά σας σχόλια ε, τους επόμενους μήνες. Να ξεκινήσω καταρχάς με τις προβληματισμούς για την αποκάλυψη των κινδύνων ε, και τις νόσεις για τις αποδόσεις κτλ. Πρώτον για τους κινδύνους. Ε, αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για τον καταναλωτή προκειμένου να πάρει την επενδυτική του απόφαση. Θέλουμε ε, ο δείκτης του κινδύνου να παρουσιάζεται στο κίνδυ και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο κίνδυνος του χύψη προϊόντος, όλα αυτά να παρουσιάζονται στο κίνδ ε, απλά. Και η απλή παρουσίαση φαίνεται ότι είναι και η καλύτερη. Τώρα, από πλευράς μεθοδολογίας, έχουμε τρεις προσεγγίσεις, προέκυψαν αυτές στο, ε, στο τεχνικό έγγραφο που δημοσιεύσαμε πρόσφατα και είναι υποσυζήτηση. Πρώτον, χρήση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και δεύτερον, χρήση μόνο ε, ποσοτικών κριτηρίων. Αναλύουμε το feedback στο έγγραφο τεχνικής συζήτησης για να ε, μειώσουμε τις επιλογές πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη ε, τα διάφορα είδη πρίψε επενδυτικών αυτών προϊόντων. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει τέλεια λύση ε, πάντοτε θα υπάρχουν ανταλλάγματα και αντισταθμίσματα που θα πρέπει να δοθούν ή να βρεθούν. Και έχουμε διαφορετικά προφίλ κινδύνου και διαφορετική εξάρτηση από τον κίνδυνο αν θέλετε. Όμως ε, αν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία ε, θα υπάρχει εμπιστοσύνη και είμαι πεπισμένος ότι οι τελικές μας προτάσεις θα είναι σημαντικό βήμα έτσι ώστε οι κίνδυνοι σε κάθε επιδετικό προϊόν να είναι όλο και πιο διαφανείς και αποκεκαλυμμένοι. Ξέρουμε ότι οι καταναλωτές συχνά δεν μπορούν να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή και ε, θα πρέπει το κόστος το ενημέρωσης να αναφέρεται επαρκώς. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις. δυσκολεύεται κανείς να αξιολογήσει την πληροφόρηση που έχει για το κόστος, το κόστος διαφορετικών προϊόντων και διαφορετικών δομών διάρθρωσης του εκάστατου προϊόντος και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με και δουλεύουμε πάνω στα RTS, καταδυστικά τεχνικά πρότυπα. Θέλουμε να έχουμε ένα summary cost indicator, ένα δείκτη ε, περιληπτικό του κόστος που θα συμπεριλαμβάνει ε, ε, τα ρητά κόστη και τα έμεσα και τα κόστη που προκύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θέλουμε το παιχνίδι να είναι επίση όρις μεταξύ των, μεταξύ των προϊόντων. Και οφείλουμε να εξετάσουμε προσεκτικά τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων προϊόντων. Από πλευράς κόστους, για παράδειγμα, έχουμε ασφαλιστικά προϊόντα και premium που έχουν να κάνουν με ε, το ε, βιομετρικό κίνδυνο. Και τέλος, Θέλω να κάνω δύο-τρία σχόλια για τις αποκαλύψεις ως προς την ενδυνάμει απόδοση κάποιου προϊόντος. Διάφορες είναι οι επιλογές για το πώς θα παρουσιάζουμε αυτή την πληροφόρηση. Π.χ. η σενάρια τι θα συνέβαινε εάν ή μια συνολική προσέγγιση ή συνδυασμό των δύο. Όσοι παρέχουν τα προϊόντα περιγράφουν λοιπόν ε, πώς θα διαμορφωθεί το προϊόν υπό διαφορετικές συνθήκες της αγοράς αλλά δεν θα δοθεί ενημέρωση ε, πιθανοτήτων του έλευσης του σενάριου του συγκεκριμένου. Η δεύτερη επιλογή τώρα είναι ε, η ενημέρωση με βάση την ε, ύπαρξη των ενδυνάμει αποδόσεων. Αυτά μπορεί να αποκαλύπτονται και να μην αποκαλύπτονται στο KIT, στο βασικό πληροφοριακό έγγραφο. Το σημαντικό είναι οι επενδυτέ να καταλάβουν ότι η ενημέρωση είναι πιθανολογική και γι' αυτό η απλούστευση στην ενημέρωση είναι καλύτερη και σε αυτό το επίπεδο των αποδόσεων και όχι μόνο στους κινδύνους. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε ο κύριος Μπαγέ έχει το λόγο. Δεν ξέρω πόσο θα μιλήσετε γιατί ο κύριος Νίντε Μάγερ πρέπει να ε, φύγει στις 6 παρα 5. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτώ τον Πρόεδρο γιατί είναι ο πιο δυνατός, ο πιο μεγάλος, ο πιο ισχυρός. Σε κάθε περίπτωση σε εσά απευθύνομαι κύριε Μάιζορ Κοιτάξτε, είναι νομοθετικό αυτό το κείμενο, το ΚΙΔ, που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναεξισορροπήσει για να έχουμε αποτελεσματική προστασία των μικροεπενδυτών και μικροπρομηθευτών ε, χρηματοπιστωτικών και χρηματιστηριακών προϊόντων που είναι περίπλοκα και συνδέονται με διαφορετικά προφίλ κινδύνου. Και ο βασικό φόβο που είχε εκφραστεί τότε από τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε να κάνει με το γεγονό ότι το KID δεν προορίζεται στην ενημέρωση των επενδυτών για να λάβουν κατάλληλη απόφαση, αλλά για να βοηθήσει ε, τους προμηθευτές να προμηθεύσουν, να πουλήσουν το προϊόν τους. Επομένως, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πτυχές που είναι απαραίτητες στην νομοθεσία αυτή, δηλαδή επιλογή ε, δικτών κινδύνου, σενάρια ε, απόδοσης και παρουσίαση διαφόρων κινδύνων που συνδέονται με το επιλεγμένο ή επιλεγέν προϊόν. Ποια προσέγγιση λοιπόν πρέπει να υιοθετήσουμε ως προς την αναδιανομή ή κατανομή των εσόδων αναλόγως με τους κινδύνους με τις αποδόσεις που συνδέονται με κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υποσημειώσει ότι δεν είναι επαρκές κριτήριο να βασίζεται κανείς σε προηγούμενες αποδόσεις για να αξιολογήσει την απόδοση και τον κίνδυνο για το μέλλον του εκάστοτε και λόγω προϊόντος, σας το υπενθυμίζω αυτό και άλλωστε όλα αυτά εξαρτώνται ε, περισσότερο από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς γιατί η τρέχουσα τιμή της αγοράς ε, σωματώνει όλους τους κινδύνους μια και έτσι ο καταναλωτής μπορεί να εξετάσει καλύτερα το κίνδυνο που συνδέεται με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό προϊόν και τις ενδυνάμει απώλειες. Λοιπόν, ε, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την προσέγγιση, για το ποια είναι τα εμπόδια που εμποδίζουν την τυποποίηση ακόμα και ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την ποιότητα της πληροφορίας που ενσωματώνεται στο KID, στο ε, βασικό πληροφοριακό έγγραφο. Κύριε Νίδερμα, σας ευχαριστώ. Μιλάω εξ ονόματος ε, του, κύριε, Πιέτη, της κυρίας οπότε μπορείτε να απευθυνθείτε τις ερωτήσεις σας ε, σε αυτήν. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Πιετικάνη να σας ευχαριστήσει για την πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά και τις αποφάσεις επίπεδο 1 αλλά και το Κοινοβούλιο. Βλέπω πως υπάρχουν τρίων ειδών κίνδυνοι, κίνδυνοι αγοράς ε, πίστης ε, και ρευστότητας και θεωρεί πως θα πρέπει όλα αυτά να υπάρχουν σε, ένα, σε μια γραφική παράσταση ή σε ένα πίνακα μαζί. Επιπλέον θεωρεί πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα του χρόνου, δηλαδή πόσο ε, το ποσό και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου, το ύψος και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου αλλάζουν σε τον χρόνο. της χάρη. Στην περίπτωση κάποιων ε, στοιχείων ενεργητικού τα οποία έχουν ε, παγιδευτεί. έπρεπε αυτά να επενδυθούν σε μία ε, πετρελαϊκή εταιρεία ή θα λαμβάνουν υπόψη και τους ε, κλιματικούς ε, κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά και τον σχεδιασμό των δικτών κινδύνου. Η ΣΥΡΠΑ επίσης θα ήθελε να ρωτήσει αν έχετε σκεφτεί καθόλου την οπτικοποίηση της σύνοψης που θα έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν κάποια πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τώρα τα σενάρια αποδοσής και το κόστος. Η κυρία Κάινεν θεωρεί πως τα σενάρια απόδοσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα σενάρια κόστους. Θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα του κόστους, το συνολικό κόστος να εμφανίζεται με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι στο δυνατόν πιο ευρύτερο. Επίσης το σωρευτικό κόστος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιληφθούν ε, οι λιανικοί επενδυτές και είναι δύσκολο βεβαίως λόγω της διαφοράς μεταξύ των τρίψ και του μέσου κόστους τους. Ε, η ΕΣΑ λοιπόν πώς θεωρεί πώς μπορούμε να το συνοψίσουμε αυτό και για τα άπαξ και για το σωρευτικό κόστος. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάιερ Η κυρία Σουίνμπορν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω εξ ονόματος ε, του Σαϊτ Καμάλ που επίσης απουσιάζει. Ε, βλέπω όμως πως απουσιάζουν και οι βουλευτές και δεν νομίζω ότι αυτό όμως σημαίνει πως υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Όμως μου έδωσε ο δόκτωρο Καμάλ κάποιες ε, σημειώσεις και πολλά από αυτά τα οποία ήθελα να πει έχουν ήδη κάλυφθει. Οπότε σας ευχαριστώ, αλλά προφανώς ο στόχος που έχουμε είναι να έχουμε ένα φιλικό έγγραφο το οποίο θα μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τα διάφορα προϊόντα. Και βεβαίως ε, το γεγονός ε, το ότι είχαμε ήδη κάποια διαβούλευση σημαίνει πως ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Εγώ θα ήθελα να δω και άλλες διαβουλεύσεις βεβαίως πριν από το τελευταίο σχέδιο και βεβαίως αυτό θα εξαρτηθεί και από τις δοκιμές που θα γίνουν με τους ε, καταναλωτές και πραγματικά μας ενθαρρύνει να ακούμε το ότι είναι χρήσιμη αυτή η διαδικασία και φαίνεται πως ήδη είχαμε κάποια χρήσιμα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν μια τελική έκθεση καθώς ε, θεωρώ πως υπάρχει κάποια αξία η οποία πηγαίνει πολύ παραπέρα από το συγκεκριμένο νομοθέτημα για να αντιληφθούμε ακριβώς το πώς ε, λαμβάνουν οι επενδυτές τις αποφάσεις. Προφανώς θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι το χρήσιμο και το συνολικό κόστος ε, που ανέφεραν ήδη οι σοσιαλδημοκράτες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης αντιλαμβάνομαι πως η διαβούλευση με τα πάνελ καταναλωτών έδειξε πως προτιμούν έναν απλό αριθμό. Αλλά δεν θα ήθελα εγώ ε, να έχουμε ένα νούμερο το οποίο θα αποκρύπτει το λεπτομερές κόστος εάν θέλει να το δει ο καταναλωτής. Γιατί βεβαίως ε, μπορεί να είναι αρκετά σημαντικό αυτό το κόστος και θα πρέπει να συγκρίνουμε παρόμοια πράγματα. Έτσι. Είτε μιλάμε για το κόστος ή τα τέλη της συναλλαγής, τέλη διαχείρισης ε, και τέλη ε, αποχώρησης. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν άλλο ένα επίπεδο πληροφόρησης εάν το απαιτήσει ο επενδυτής. Και εδώ μιλάμε για την MIFID και τη σχέση της με αυτό το θέμα. Η MIFID απαιτεί νομίζω τα, το κόστος συναλλαγής να είναι το ελάχιστο δυνατό, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε ένα νούμερο το οποίο θα κρίνει και την ορθή εκτέλεση στο μέλλον. Οπότε με καθυσίχασε ο κύριος Μαγιόρ που είπε ότι θα προσπαθήσει να συντονιστεί με την ΜΥΦΙΔ όσον αφορά την ΠΡΙΠΣ την οδηγία αυτή εδώ. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το έβρος των προϊόντων που καλύπτονται. Και τέλος το τελευταίο ερώτημα του δόκτρος Καμάλ μιλήσατε για κατηγορίες κινδύνου και αυτός υπέθεσε ότι θα βασίζονταν στα εργαλεία του usage και θα ήταν κάτι το ανάλογο. Αυτό χρειάζεται όχι μόνο για να το αντιληφθούν οι επενδυτές αλλά και για να μην είναι υπερβολικό το βάρος για αυτούς που θα φτιάχνουν αυτά τα προϊόντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Σουίνμπορν κύριος Γκίγκολτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να περιοριστώ σε πράγματα που δεν ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη δουλειά που κάνατε εδώ πέρα. Και τώρα ένα έγγραφο τριών σελίδων χρειάζεται 160 σελίδες για να καλύψει δύο μόνο από τα ζητήματα που προέκυψαν, κάτι το οποίο αποκαλύπτει πως είναι δύσκολο τα απλά πράγματα να γίνουν σύντομα και μπορούμε να διαστευλώσουμε τις αγορές. Από την άλλη είναι μια τεράστια ευκαιρία να βρεθούν πάρα πολλά άσχημα προϊόντα στην αγορά. Οπότε, για τις διάφορες επιλογές ε, τώρα θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. μια επιλογή ήταν ε, το Τζάιλ, μια άλλη ήταν ε, αυτή η απόδοση την οποία αναφέρεται και το κόστος ως ποσοστό να δεν ξέρω αν προστατεύεται έτσι ο καταναλωτής. Μήπως έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι πιο απλό. Δηλαδή να μιλήσετε για μείωση του πλούτου. Γιατί αυτό το αντιλαμβάνονται ευκολότερα οι περισσότεροι καταναλωτές σε σχέση με την πιθανή απόδοση. Και επίσης ε, νομίζω πως ε, Δεύτερον, τώρα μιλάμε για τους ε, κινδύνους και το τι βεβαίως παίρνει κανείς σε αντάλλαγμα. Ένα πράγμα το οποίο λείπει βεβαίως είναι ένα σενάριο απόδοσης και το τι υποθέσεις έχουν γίνει για να βγει αυτό το σενάριο. Τα σενάρια αυτά βεβαίως είναι κάπως ε, δύσκολα πράγματα και θα ήθελα να γνωρίζω πώς θα διασφαλίσετε την συγκρισιμότητα των ε, διαφόρων αυτών σεναρίων που συντάσσουν η παραγωγή αυτών των προϊόντων. Ποια θα είναι τα τυποποιημένα κριτήρια για να φροντίσετε ε, δεν ξέρω γιατί γελάει η Κομισιόν. Πού είναι το αστείο. Ποια θα είναι λοιπόν τα τυποποιημένα κριτήρια και πώς θα διασφαλίσετε ότι θα λειτουργούν. Τώρα, όσον αφορά τους κινδύνους. Κάνετε κάποιες δοκιμές όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας ε, και πίστης και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Και τέλος, να τονίσω πως ε, βλέπω πως ε, είδατε δύο από τα βασικά ε, ζητήματα και βλέπουμε εκεί πέρα πως ε, το όλο ζήτημα των βιώσιμων επενδύσεων ε, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε ολόκληρο το Κοινοβούλιο, δηλαδή να έχουμε κάποια στιβαρά κριτήρια για να λέμε ότι κάτι είναι το βιώσιμο και από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πολύ ε, δουλειά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω εγώ από την Κομισιόν και τους πολιτές αυτών των προϊόντων να ξεκινήσουν βεβαίως να ασχολούνται με αυτό το θέμα όταν τους ανατεθεί αλλά νομίζω πως ε, για να σταματήσει αυτό το πράσινο ξέπλυμα αφενός και να ενθαρρύνουμε την αγορά αφετέρου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκίγκολτ. Θα δώσουμε τον λόγο τώρα πρώτα απ' όλα στην Κομισιόν στον κύριο Γκέντερ. Um, Αν κατάλαβα καλά, εγώ κυρίως θα απαντήσω στις τελευταίες ερωτήσεις που αφορούν το αποτέλεσμα για τα κόστη και την επιστροφή απόδοσης. Η μελέτη καταναλωτή ε, έδειξε βασικά ότι τα βάση, τα, τα διάφορα μέτρα, οι διάφορες μετρήσεις δεν είναι ευνόητες. Δεν υπάρχει σαφές αποτέλεσμα για το κατά πόσο είναι επιστροφή απόδοση ή άλλοι δείκτες που είναι προτιμότεροι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο ει βάθος και όπου απλώ πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε το καλύτερο αποτέλεσμα μαζί με τις ΕΖΑ. Τώρα, τα σενάρια απόδοσης θα τα αφήσω στο κύριο ε, στο Στίβεν, γιατί αυτό έχει συζητηθεί σε επίπεδο μεικτή ΕΖΑ για τις επενδύσεις Υπάρχει κάτι στο προηγούμενο κείμενο και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, ε, το έχουμε ήδη συζητήσει. Ε, βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα ήδη από τώρα να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με αυτό και φυσικά θα πρέπει να το ακολουθήσουμε και να το προπτεύσουμε σωστά. Αυτή τη στιγμή όπως σας είπα το παρακολουθούμε και βέβαια Έχουμε υπόψη μας και τη ρήτρα αναθεώρησης, αλλά βεβαίως δέχομαι τα όσα είπατε, για τα όσα μπορεί να χρειαστεί να γίνουν σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέρνερα και τέλος το λόγο έχει ο κύριος Μέιζορ. Κάποιες οι πρώτες γενικές παρατηρήσεις και έπειτα θα δώσω το λόγο στον Τιμ, αν συμφωνείτε κι εσείς. Καταρχήν, το KIT θα πρέπει να είναι ένα ε, έγγραφο που θα ενημερώνει τον, τον επενδυτή ε, και δεν θα είναι το ίδιο το προϊόν. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι από το γεγονός ότι οι επενδυτές δεν καταλαβαίνουν ακριβώς το προϊόν στο οποίο επενδύουν και γι' αυτό και θα πρέπει να ε, ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές ώστε να μπορούν σωστά να λάβουν τις αποφάσεις τους εν πλήρη γνώση του θέματος. Ε, τώρα, τα σχόλιά σας θα τα λάβουμε υπόψη στην υπεραιτέρω εργασία μας και αναφέρονται στο, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, δηλαδή να απλοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να ομαδοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να είναι κατανοητό. Ενώ από την άλλη πλευρά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο περισσότερο ομαδοποιούμε, πολύ σημαντικές πληροφορίες χάνονται και άρα εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Υπάρχει το παράδειγμα για τους κινδύνους. Ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεκάθαρος δείκτης κινδύνου και μετά αρχίζουμε ε, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αγοράς και ούτω καθεξής. Τώρα, ανάλογα με τις επενδυτικές προτιμήσεις καθενός, αξιολογεί διαφορετικά το προϊόν με βάση τους ε, κινδύνους που εμπεριέχει. Το ίδιο και για το στοιχείο του κόστους. Πώς αυτό το ομαδοποιούμε. Το κόστος δηλαδή του στοιχείου ασφάλισης είναι πολύ διαφορετικό από άλλα κόστη που σχετίζονται με το προϊόν. Από τη μια πλευρά θέλουμε να δώσουμε μια ομαδοποιημένη και συνολική εικόνα γιατί θα καταλάβει τι πρέπει να πληρώσει, αλλά από την άλλη πλευρά θέλεις να δώσεις και τις απαραίτητες πληροφορίες. Εάν δηλαδή το κόστος είναι διαφορετικής φύσης, είναι διαφορετικό από το κόστος της ίδιας της ασφάλισης. Προτίμηση λοιπόν προς την απλοποίηση από τη μια πλευρά και την ε, ε, ομαδοποίηση την, ε, την παρουσίαση ενός συνολικού προϊόντος, από την άλλη πλευρά να μην χαθούν οι σημαντικές πληροφορίες για τον επενδυτή. Τώρα, σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών, αυτό είναι ο στόχο του Νοεμβρίου. Ο σχεδιασμός, το σχέδιο δηλαδή τεχνικών προδιαγραφών πριν ολοκληρώσουμε το Μάρτιο του επόμενου έτου, πολύ σύντομα για τη διαδικασία δηλαδή. Για το θέμα του ε, πεδίου εφαρμογή, ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε, τα νομικά ζητήματα, είναι η συμπερίληψη ή όχι των παραγόγων. Υπάρχουν θέματα για το πεδίο εφαρμογή και ξεκολουθούμε να τα εξετάζουμε και είναι σωστό να σας πω ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτή η συζήτηση σε σχέση με τα παράγωγα, για παράδειγμα. Το θέμα τώρα της βιωσιμότητας. Βεβαίως η βιωσιμότητα θα είναι ένας δείκτης, ένα ενημερωτικό στοιχείο στο ίδιο το πακέτο. Το θέμα είναι πότε μπορεί κανείς να πει ότι είναι βιώσιμο το προϊόν. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εντολή και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να ε, συντονιστούμε με την Επιτροπή και να δουλέψουμε για αυτή την ιδέα, για το πώς δηλαδή αξιολογεί κανείς κατά πόσο μια, ένας ισχυρισμός βιωσιμότητας είναι ε, δικαιολογημένος. Τέλος, ε, για τη συζήτηση για το TCR, τη μείωση απόδοσης, για να χρησιμοποιήσω και αυτή τη δύσκολη λέξη, η μείωση απόδοση είναι μεγαλύτερη από τη μέτρηση του, συνολικού κόστου γιατί λαμβάνει υπόψη καλύτερα τις χρονικέ διαφορές, τη διάρκεια ζωή του προϊόντος, αλλά βέβαια δεν έχουμε ακόμα τελική θέση από αυτό. Δύο λεπτά ακόμα ώστε ο Τίμ να ολοκληρώσει τη δική μα συμβολή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ναι, συγγνώμη, ναι, βεβαίω μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύψατε πολλά από τα θέματα που μπορούμε να αναπτύξουμε σήμερα το απόγευμα. Το σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ή μάλλον να το πω αλλιώς. Ε, δεν μας εκπλήσει το ότι υπάρχουν 100 σελίδες για κάθε σελίδα του βασικού πληροφοριακού εγγράφου. Γιατί αυτό που προσπαθούμε να αναλύσουμε είναι κάτι το τελείως καινούριο. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι τόσο ευρύβη στο παρελθόν. Μια τέτοια προσπάθεια, μια δίκαια προσπάθεια να μπορούν να συγκριθούν τα κόστη μεταξύ των διαφόρων ε, δομών, των διαφόρων προϊόντων. Και αυτό δείχνει τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας. Τώρα, ως προς τα σενάρια ε, αποδόσεων, η σωστή στάθμιση, ο βαθμός συνταγογράφησης, αν θέλετε, ε, Πού βρίσκεται η απώλεια και η ευθύνη ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση γιατί είναι νέα προϊόντα, υπάρχει μεγάλη καινοτομία και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε με αυτό το εργαλείο να διαβάσουμε όλο, όλη την προϊόντική γκάμα και είναι δύσκολο να βρεθεί το σημείο ισορροπίας. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι το υψηλότερο επίπεδο προδιαγραφών σαφήνειας ε, του ουδέτερου σενάριου, του θετικού σενάριου ή του αρνητικού σενάριου και το καθεξής είναι στοιχεία εξαιρετικά σημαντικά. Αυτές είναι οι προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν σχόλια από τους συναδέλφους και άρα αυτή τη στιγμή γίνεται αξιολόγηση ε, του feedback σε σχέση με τα RTS που πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2016. Σήμερα λοιπόν εδώ ολοκληρώνουμε την εξέταση της σημερινής μας ημερησίας διάταξης. Αύριο θα συνεχίσουμε στις 9 το πρωί και θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης δραστηριοτήτων και εποπτείας ε, των ε, σχετικών αρχών